Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μπορούμε να αρχίσουμε νομίζω. Καλώς ήρθατε στην σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικής Ανάπτυξης, Δημοσιονομικών και Εμπορίου της ε, Κοινής Συνέλευσης ΑΚΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμπροεδρεύω εδώ με τον κύριο Τσολαπόζο μαζί τη συνεδρίαση αυτή. Εγώ θα προδρέψω τα 8 πρώτα σημεία της ημερήσιας διάταξης που θα εξετάσουμε σήμερα και η κυρία Λαμπόσο αύριο θα προδρέψει τα σημεία 9 μέχρι και 14. Για τη Γερμανία μπορείτε να μιλήσετε και να ακούσετε αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά και ελληνικά. Επιπλέον έχουμε παθητική διερμηνία στα πορτογαλικά, σημαίνει ότι μπορείτε να μιλήσετε πορτογαλικά. Να ξέρετε ότι μέσω διαδικτύου μεταδίδεται η συνεδρίαση. Όσοι ενδιαφέρονται λοιπόν μπορούν να παρακολουθήσουν τη συνεδρίασή μας. Έτσι και άλλοι βουλευτές αλλά και ερευνητέ, φοιτητέ, διεθνείς οργανώσεις κλπ. μέλη της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να παρακολουθήσουν το έργο της συνελευσής Και τώρα θα περάσουμε στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Και το πρώτο σημείο είναι η έγκριση των... της ημερήσιας διάταξης. Είναι στους φακέλους σας. Αν δεν έχετε σχόλια ή τροποποίησεις να προτείνετε, θεωρείτε εγκεκριμένη. Συμφωνείτε? Έχετε σχόλια μήπως? Καλώς. Εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Δεύτερο σημείο. Έγκριση των πρακτικών τη τελευταία συνεδριασή μα τη 17η Δεκεμβρίου 2016 στο Ναϊρόμπι τη Κένια. Τα πρακτικά αυτά βρίσκονται στους φακέλους σας. Αν δεν έχετε να προτείνετε κάποια τροποποίηση μέχρι αύριο στις 10 το πρωί, θα θεωρηθούν εγκεκριμένα τα πρακτικά αυτά. Τρίτο σημείο. ανακοινώσει. Πριν μπούμε δηλαδή στα ουσιώδη σημεία τη ημερήσια διάταξη, θέλω να σα ενημερώσω για το εξή. Αποφάσει που έλαβε το Προεδρείο στην 33η Σύνοδο της Κοινή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΑΚΕ Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 33η η 33 η συνοδος θα λάβει χώρα στο Σεντ Τζούλιαν στη Μάλτα 19 με 21 Ιουνίου. το Προεδρείο αποφάσισε δύο θέματα για ψηφίσματα κατεπήγοντος. Το ένα είναι η κατάσταση ασφάλειας στην περιοχή Σαχέλ Σαχάρα και το δεύτερο θέμα είναι η κατάσταση στο Μπορούντι. Η προθεσμία είναι η 3η 16η Μαΐου 2017 στις 12 το μεσημέρι για την υποβολή ψηφισμάτων κατεπήγοντος. Τα δύο θέματα αυτά θα επιβεβαιωθούν βέβαια αργότερα. Επίση, το Περιτρίο αποφάσισε να οργανώσει τι εξή ε, συζητήσει. Συζήτηση κλειδί για τη δημογραφική ανάπτυξη, προκλήσει και ευκαιρίε. Πρώτο θέμα για συζήτηση χωρί ε, ψήφισμα θα είναι ο κίνδυνος της ε, ανάδυσης μιας πιο σοβαρή ε, πείνα λοιμού και ανθρωπιστικής κρίσης στην ιστορία. Δεύτερο θέμα συζήτησης χωρίς ψήφισμα είναι η μετανάστευση, κατάσταση πραγμάτων και η προθεσμία για να υποβληθούν ερωτήσεις για προφορική απάντηση από την Επιτροπή και το Συμβούλιο είναι η Παρασκευή 31 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι. Η περιφερειακή συνάντηση για τον ειρηνικό θα λάβει χώρο στο Βανουάτου 19 με 21 Ιουλίου 2017. Όσον αφορά το newsletter, παρουσιάζει τα αποτελέσματα της συνάντησής μας στο Ναϊρόμπι 19 με 21 Δεκεμβρίου 2016 και υπάρχει στα γαλλικά και στα αγγλικά στην είσοδο της αίθουσάς μας. Επίσης υπάρχει το newsletter και σε ηλεκτρονική μορφή. Αν θέλετε να το παίρνετε αυτόματα, στείλτε ένα αίτημα με email στη διεύθυνση acp.europar.europa.eu. Και τώρα, η Συμπρόεδρος να μας πει αν έχει και εκείνη να κάνει ανακοινώσεις, παρακαλώ. Όχι. Καλώς. Συνεπώς μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης τώρα. Το τέταρτο σημείο λοιπόν είναι οι επιπτώσεις του διεθνούς εμπορίου και της πολιτικής εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά στην ε, αλυσίδα αξιών. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι η σύλληψη, ο σχεδιασμός και η παραγωγή των προϊόντων αποτελούν σημαντικά βήματα και λαμβάνουν χώρα σε διάφορα σημεία. οι δασμοί έχουν λιγότερη σημασία από ό,τι είχαν κατά το παρελθόν. Οι εισαγωγέ ε, ανταλλακτικών αποτελούν όλο και πιο σημαντικό κομμάτι των εμπορικών συναλλαγών. Οι δασμοί και η χώρα προέλευσης λοιπόν αποκτούν νέα σημασία. Η κυρία Ρένα, η εισηγήτριά μας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν είναι εδώ, οπότε ίσως να την περιμένουμε να περάσουμε στο πέμπτο σημείο και μετά να πάμε πίσω στο τέταρτο όταν θα είναι εδώ. Λυπάμαι. Γι' αυτό. Ίσως έχει ανελημμένες υποχρεώσεις ταυτόχρονα και να αργήσει λίγο. Λοιπόν, σημείο 5 βελτίωση της ε, βοήθειας και της ε, αποτελεσματικότητας των αναπτυξιακών μας προσπαθειών. Οι συγητέ είναι ο Σεμπάστιαν Καπουλάντα και ο Νεοκλής Σιλικόδης που έχουν ετοιμάσει ένα σχέδιο έκθεση που θα συζητήσουμε σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω και του δύο συνεισηγητέ για το έργο του και του παρακαλώ να μα παρουσιάσουν την έκθεσή τους για την αποτελεσματικότητα αυτή της ε, βοήθειας και των αμυσιακών μας προσπαθειών είναι κάτι πολύ σημαντικό για την κυριαρχία των χωρών δικαιούχων και χρειάζεται συγκεκριμένες διαδικασίες. Όχι δάνεια, αλλά επιχορηγήσεις. Θα δώσω λοιπόν το λόγο πρώτα απ' όλα στον Σεμπάστιαν Κοπουλάντα, έναν από τους δύο εισηγητές. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Συμπρόεδρε. Σας ευχαριστώ και τις δύο πρόεδρους. Κυρία Πρόεδρε, ήδη ευθύς εξ αρχής θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον συνεισηγητή μου που βοήθησε να συντάξουμε το κείμενο αυτό και τα συνοδεύοντα ψηφίσματα. Χαίρομαι που παρουσιάζω την έκθεση αυτή. Να ξέρετε ότι είμαστε έτοιμοι και με τα ε, ψηφίσματα τα οποία θα εγκριθούν τον Μάλτιο, το, στη Μάλτα τον Ιούνιο. Αναφέρονται πολλά ζητήματα στα ψηφίσματα που καλείται να εξετάσει το σώμα μας για να διασφαλίσουμε ότι η συνεργασία μεταξύ των ε, περιοχών μας πετυχάνει τους στόχους που είναι η βοήθεια στην ανάπτυξη και την μείωση της ένδυας στις χώρες δικαιούχους. Κύριε Πρόεδρε, η αναπτυξιακή βοήθεια προσφέρεται και για την ανάπτυξη υποδομών, για προγράμματα για την πραγματική οικονομία, τον κοινωνικό τομέα, δημοσιονομική στήριξη και προγραμματική βοήθεια επίσης. Παρ' όλα αυτά, το σχέδιο έκθεσης που έχουμε μπροστά μας εκφράζει την δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν κατάφερε να πετύχει το 0,7% του έψη αναπτυξιακή βοήθεια από τις χώρες μέλη. Σήμερα είμαστε στο 0,47%. Η αποτυχία αυτή, κυρία Πρόεδρε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταποκριθεί στους στόχους που έθεσε για το 2015 σημαίνει πάνω από 2 δισεκατομμύρια αμερικανικά δολάρια, τα οποία δεν πήγαν τελικά στις υποανάπτυξη χώρες για να πετύχουν τους στόχους της χιλιετίας. Η έκθεση λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, λέει ότι το θέμα αυτό απαιτεί άμεση προσοχή από τις χώρες μέλη, προκειμένου οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης να επιτευχθούν μέχρι το 2030. Επιπλέον, η έκθεση υπογραμμίζει και την ανάγκη που υπάρχει να στηρίξουμε την εκπαίδευση για να υπάρξει βιωσιμότητα μακροπρόθεσμα και αποτελεσματικότητα των προσπαθειών. Η έκθεση λέει επίσης ότι οι επιπτώσεις της βοήθειας, ο αντίκτυπος της βοήθειας δεν ήταν αυτός που περιμέναμε σε ένα μεγάλο βαθμό επειδή οι δωρητές προσπαθούσαν να πετύχουν τους δικούς τους στόχους και τις δικές τους προτεραιότητες στις χώρες δικαιούχους. Οπότε η έκθεση και τα συνοδεύοντα ψηφίσματα ζητούν αλλαγή στην προσέγγιση αυτή. Κύριε Πρόεδρε, ο ιδιωτικός τομέας και η συμμετοχή του για επενδύσεις προς τις χώρες ΑΚΕ πρέπει να επιταχυνθεί. Και αυτό για να υπάρξει δημιουργία θέσεων απασχόλησης που θα εξασφαλίσουν βιώσιμη ανάπτυξη. Κύριε Πρόεδρε, θα θέλαμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου οι χώρες δικαιούχοι να έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τη βοήθεια που τους προσφέρεται να μην ε, ξεχνώνται και να συμμετέχουν και στις επενδύσεις και στο εμπόριο. Τα ψηφίσματα, κυρία Πρόεδρε, και η έκθεση μεταξύ άλλων λένε τα εξής. Έχει μεγάλη σημασία το τι θα αποφασίσουν οι ίδιες χώρες και η κυριαρχία των ίδιων αυτών των χωρών δικαιούχων και τονίζει ότι η ευρωπαϊκή βοήθεια δεν θα πρέπει να βασίστε στις προτεραιότητες των δόρυτων, αλλά να προσαρμόσετε με τους στόχους των χωρών δικαιούχων. Δεύτερον, υπογραμμίζει και ζητάει πιο προσεκτική αξιολόγηση των τοπικών αναγκών από τους δωρητές, έτσι ώστε η βοήθεια να είναι όσο γίνεται πιο πολύ αποτελεσματική και η βοήθεια αυτή να δίνεται έγκαιρα και σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέγουν βάσει μηχανισμών που θα διασφαλίζουν επίσης ότι η βοήθεια που πηγαίνει στις χώρες δικαιούχους θα χρησιμοποιείται αποτελεσματικά. Το ψήφισμα ζητάει από τις χώρες να καθορίσουν αναπτυξιακές προτεραιότητες και σχέδια που θέλουν να εφαρμόσουν δικαιούχες χώρες. Γι' αυτό λοιπόν ζητούμε από τις χώρες μέλη να προωθήσουν ένα χάρτη πορείας για το πώς θα πετύχουν τον στόχο αυτό του 0,7% του ΕΠ από κάθε χώρα αλλά και συνολικά μέχρι το 2030 ώστε να βοηθούν οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Επιτρέψτε μου τώρα να Σα ζητήσω να εξετάσετε την έκθεση και αν έχετε τροπολογίες να τις υποβάλλετε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κοπουλάντε. Ο κύριος Ηλικιώτης Δυστυχώς δεν έχει φτάσει ακόμη στην αίθουσα, ούτε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται εδώ. Άρα θα επιστρέψουμε στο 4 σημείο της μέσης διάταξης και μετά θα ξαναπεράσουμε στο 5. Εντάξει, ξέρω ότι δεν είναι και καλύτερη δυνατή διαδικασία αυτή, αλλά τέλος πάντων. Να περάσουμε στο σημείο 4 λοιπόν της μέσης διάταξης που είναι ο αντίκτυπο ε, το διεθνού και των εμπορικών πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Παγκόσμια Αλυσίδα Αξία. Σα είπα ότι το 70% του παγκόσμιου ΑΕ παράγεται μέσω παγκόσμιων αλυσίδων αξία, που σημαίνει ότι η σύλληψη, ο σχεδιασμό, δηλαδή η μελέτη, η παραγωγή προϊόντων γίνεται με μια σειρά σταδίων σε πολλές χώρες. Αυτό επηρεάζει την εμπορική πολιτική. Οι εισαγωγικοί θεσμοί έχουν λιγότερη, μάλλον, λιγότερη σημασία από τη διάκριση μεταξύ, από ό,τι παλιότερα λόγω του ότι δεν είναι σαφής η διάκριση μεταξύ εισαγωγών εξαγωγών, εισαγωγέ ανταλλακτικών, όπω που τις εξαγωγές στη συνέχεια ε, συντάσσονται όλο και περισσότερο στις εμπορικές ε, ροές. Ε, τα εισαγωγικοί δασμοί και οι προέλευση. επομένως, έχουν μια διαφορετική σημασία. Πρέπει να προσαρμόσουμε τι πολιτικές μας περί πρέπει να είμαστε πιο ανοιχτοί στο εμπόριο. Αυτή είναι η απάντηση. Αυτό όμω πώ θα επηρεάσει τι αναπτυσσόμενε χώρε και πώ θα φροντίσουμε τη ρύθμιση των ε, παγκόσμιων εταιριών. Ε, η συγκέντρια ε, για τον αντίκτυπο του διεθνούς εμπορίου και των πολιτικών, εμπορικών πολιτικών της Ένωσης Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας είναι η Μαρία Ρενά. Και από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου μας λέει ποιες είναι ε, προκλήσει τα βασικά θέματα θα σας ε, φανεί σίγουρα ενδιαφέρον το θέμα. Θα ζητήσω από την κυρία Ρενά να κάνει μια σύντομη παρουσίαση. Έχετε και το έγγραφο εργασία σα στο φακέλο σα. Παρακαλώ κυρία Ρενά. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι, είμαι αρμόδια στο πλαίσιο τη Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου για την κατάρτιση έκθεση με τίτλο «Τον αντίκτυπο της διεθνούς, ε, τον του Διεθνούς Εμπορίου και των Εμπορικών Πολιτικών της Ένωσης Παγκόσμιας Αλυσίδας Αξίας. Αποφάσισε η Ένωση να συντάξει τη σχετική έκθεση, γιατί έπρεπε να προβληματιστούμε πάνω στον τρόπο με τον οποίο μπορεί εμπόριο και επενδύσεις να βελτιώσουν ε, τις ε, παγκόσμιες αλυσίδες αξιών, που να είναι πραγματικά εργαλεία, που θα υπηρετούν την οικονομία αλλά όχι μόνο απλά την οικονομία, τη βιώσιμη, αηφόρη οικονομία και για την Ευρώπη και για τους εταίρους της. Ε, και αυτές οι αλυσίδες αξίας είναι ένα σημείο κλειδί της παγκόσμιας οικονομίας είναι στο επίκεντρο των εμπορικών και επενδυτικών πολιτικών. Η διεθνής παραγωγή διαρθρώνεται κυρίως γύρω από παγκόσμιες αλυσίδες αξιών και στις περισσότερες περιπτώσεις πολυεθνικές ε, συντονίζουν μέσω των διασυνδεδεμένων θηγατρικών εταιριών ε, ή από ανεξάρτητους προμηθευτές ε, ή από μεμονωμένους συνεργαζόμενους φορείς που μπορεί να εργάζονται και στην άτυπη Άρα δεν υπάρχει επαρκής προστασία. Σήμερα τα τελικά προϊόντα είναι γύρω στο 25% του παγκόσμιου εμπορίου. Βλέπουμε λοιπόν ότι είτε οι πόροι είτε τα συστατικά μέρη, ανταλλακτικά κτλ. των τελικών προϊόντων είναι τα βασικά αγαθά. Έχουμε το commerce for all, το εμπόριο για όλους, ε, trade for all. Είναι μια στρατηγική εμπορική αυτή, με στόχο μια επενδυτική εμπορική πολιτική που θα είναι πιο υπεύθυνη Υποτίθεται ότι θα πρέπει και λέω ότι πρέπει να είναι υπεύθυνη. Εδώ βλέπετε και κάποιους περιορισμούς δηλαδή. Ο στόχος επίσης είναι και όλη η αλυσίδα να γίνει πιο υπεύθυνη. Θα ήταν λίγο παράλογο λοιπόν να είναι λόγω υπεύθυνο μόνο το ευρωπαϊκό σκέλος, αν δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει υπευθυνότητα και ευθύνη για όλη την αλυσίδα. Και με την προσπάθειά μας για την καταπολέμηση φοροαποφυγής, ε, παρελθόν των πολυεθνικών. Είπαμε ότι χρειάζεται να έχουμε πολιτικές διαφάνειας, δεούσας επιμέλειας, ε, στην αλυσίδα εφοδιασμού και κοινωνική εταιρική ευθύνη και περιβαλλοντική ε, εταιρική ευθύνη. Έχει κάνει συστάσεις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά στρατηγική. Τονίζουμε την ανάγκη να είναι υποχρεωτικά τα κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη που προβλέπονται σε όλες τις συμφωνίες ε, ελευθέρων συναλλαγών που συνάπτει η Ένωση με του εταίρου τη. Επίση ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια διπλή προσέγγιση. Αφενό, να διαφυλάξουμε δηλαδή τα κοινωνικά περιβαλλοντικά μοντέλα, αλλά ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη και αξιοπρεπή θέση εργασία για την απασχόληση και για τι χώρε εταίρου. Το Κοινοβούλιο καλεί επίση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει τη δέουσα επιμέλεια, όπω ε, αυτό θεσπίζεται σε επίπεδο όσα. Πρόσφατα εγκρίθηκε ένας κανονισμός ε, για τα μεταλλεύματα από χώρε σε εμπόλεμη κατάσταση. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εμείς πρέπει ε, να δούμε και την εθελοντική διάσταση ε, που θέλουμε να γίνει δεσμευτική σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο τομέα. Η εμπορική πολιτική σε διάφορους τομείς επικρίνεται έντονα όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά κυρίως στην Ευρώπη και στο πλαίσιο της περιφερειακής ε, συνέλευσης αυτά. Συζητήσαμε πολύ τις εμπορικές συμφωνίες, ε, εμπορικές και οικονομικές συμφωνίες. Βλέπουμε ότι ιδίω στην Αφρική και των πολιτών ανησυχεί με αυτές τις συμφωνίες ε, ελεύθερων συναλλαγών. Η απάντηση που πρέπει να δώσουμε σίγουρα δεν πρέπει να είναι μια προστατευτική απάντηση. σαν αυτή ε, του προγράμματος του Πρόεδρου Τραμπ. Αντίθετα, πρέπει να ε, προτάσεις πάνω στις αξίες του εμπόριου. Θέλουμε λοιπόν η παγκοσμιοποίηση να είναι πιο δίκαιη, πιο διαφανής και ευθυγραμμισμένη με τις προκλήσεις της εποχής μας. Ιδίω δηλαδή θεματολόγια 2030 για μια βιώσιμη ανάπτυξη για όλους. Είναι σημαντικό λοιπόν να τα ζητήματα της υπευθυνότητα, της διαφάνειας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της φορολογικής δικαιοσύνης, της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης, να τα βάλουμε στο επίκεντρο του κοινοβουλευτικού μας έργου, να δείξουμε στους Ευρωπαίους πολίτες πως το εμπόριο μπορεί να είναι μοχλός για μια πιο δίκαιη παγκοσμιοποίηση και με αυτό το πνεύμα έχω εκπονήσει ένα γράφο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο θα συζητήσουμε εδώ, γιατί είναι ένα κοινό έγγραφο εργασία ε, για ε, τι παγκόσμια αλυσίδε αξία, το ρόλο του στην παγκόσμια οικονομία, τι πρωτοβουλίε στο πλαίσιο τη ε, διαφάνεια και τη ευθύνη. Παραδείγματο χάρη, έχουμε το σύμφωνο δεσμότητα για τον Μπαγκλαντέ, αυτό που σα είπαμε, τα μεταλλεύματα από διάφορε πόλεμε περιοχέ, οι αρχέ των νομέθων και διάφορα άλλα μέσα. Θέλουμε επίσης να προωθήσουμε την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και των υποδομών, να μειώσουμε το κόστος του εμπορίου και των επενδύσεων που ε, αυξάνεται λόγω των ε, φιλελεύθερων πολιτικών και την ε, πρόθεση μόνο αυτήν εργατικού δυναμικού και πρέπει να δούμε και τι γίνεται με την οικονομία της Κίνας και της Ινδίας. Ε, αυτές οι αλυσίδε αξίας ε, δεν αναπτύσσονται όμορφα ανά τον κόσμο. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ε, βιομηχανισμένων χωρών, αναδυόμενων οικονομιών και φτωχότερων χωρών. Αυτά δημιουργούν αποκλήσει και ανισότητες. Και ό,τι αφορά το dumping πρέπει να το καταπολεμήσουμε και αυτό. Ο ρόλος των πολυεθνικών είναι κεντρικός. Το 50% του εμπορίου αγαθών γίνεται μεταξύ διαμεσολαβητών μέσω μάλλον ενδιαμέσων διαμεσολαβητών, ίσως από τον ίδιο πολυεθνικό όμιλο πολλές φορές. Επίσης ε, έχουμε στο έγγραφό μας βασικές προκλήσεις ε, για αυτή την διακυβέρνηση σε επίπεδο εταιρείων, κρατών και εμπορικής πολιτικής. Αναφέρουμε επίσης τι ευκαιρίες αλλά και τι ε, κινδύνους μπορεί να ενέχουν όλα αυτά. Θέλουμε να μειώσουμε τους δασμούς, έχουμε τον, τους κανόνες καταγωγής, την εμπορική διευκόλυνση, το θέμα ε, της διάστασης του φύλου, εμπορικές προτιμήσεις, ε, βιώσιμη ανάπτυξη, το αυτό το κεφάλαιο στις ε, εμπορικές συμφωνίες. Τέλος, προτείνουμε και κάποιες συστάσεις είναι στο εγγραφωμένο, αλλά μπορούμε να τη συζητήσουμε ε, και εδώ. Θεωρώ ότι η ευθύνη ε, πρέπει να καλύπτει το σύνολο της αλυσίδας, η υπευθυνότητα. Δηλαδή να ε, υπάρχει σεβασμός από όλους προς όλους και να υπάρχει δίκαιος επιμερισμός πολύ πιο ισορροπημένος του πλούτου σε σχέση με αυτό που βλέπουμε σήμερα. Ευχαριστώ. Thank you very much, Miss Arena. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Αρένα. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στα μέλη που το επιθυμούν για ερωτήσεις, σχόλια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ τον, ε, ε, την εισηγήτρια για την, ε, για την εισήγηση της. Είναι αλήθεια ότι στις αναπτυσσόμενες οικονομίες έχουν αυξηθεί ευκαιρίες ώστε να μπει κανείς σε ενδιάμεσες δυνατότητες με μικρά ποσά που προσθέτουν αξία σε οποιοδήποτε προϊόν. Είμαστε την, της άποψης ότι έχουν έτσι ανοίξει δυνατότητες για ανάπτυξη που παλιότερα δεν υπήρχαν στην παγκόσμια οικονομία. Οι αναπτυσσόμενες χώρες μπορούν έτσι τώρα να ασχοληθούν με ένα προϊόν το οποίο δίνει συγκεκριμένη προστιθέμενη αξία εφόσον ε, κομμάτια της αλυσίδας παραγωγής ανατίθεται σε εξωτερικούς συνεργάτες. Έχουμε φτάσει έτσι σε μια κατάσταση το διεθνές εμπόριο όπου το, ε, αυτό γίνεται από ενδιάμεσες ε, υπηρεσίες λόγω της δυνατότητας να καλύψουμε μόνο ένα είδος ε, δραστηριότητας υπηρεσίας, παροχής υπηρεσιών ακόμα και μικρές οικονομίες όπως οι δικές μας πρέπει να τοποθετηθούν σε ε, συγκεκριμένες αγορές. πρόκληση παραμένει ότι οι η πολιτικές είναι αυτές οι οποίες επηρεάζουν την επιτυχία των κοινοπραξιών ε, εξαρτώνται από την φορολόγηση των ε, επενδύσεων, από την αρχική ανάπτυξη, την συμμόρφωση προς τα διεθνή στάνταρ και το ευρύτερο επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο προωθεί και ευνοεί την επιχειρηματικότητα. Όλα αυτά από κοινού θα πρέπει να συνδυαστούν για να αναλύσουμε, να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε μεταρρυθμίσεις που θα επιτρέπουν την συμμετοχή ε, των κοινοπραξιών. Τώρα, δυστυχώς, λίγες είναι οι χώρες εκεί που έχουν τέτοιου είδους στρατηγικές. Πολλές εξ αυτών έχουν ε, διάφορα εθνικά σχέδια, αλλά ε, που αφορούν τις επενδύσεις ή τα σχολεία, την παιδεία. Είναι πολύ μεγάλη πρόκληση λοιπόν να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε, αυτή, σε αυτές τις ευκαιρίες. Άλλα σχόλια. So, uh, I would like to give the ε, θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον κύριο Χέντρεσον. Παρακαλώ. Κυρία Συμπρόεδρε, αξιότιμοι κυρίε και κύριοι βουλευτέ, σα ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω για αυτή την έκθεση και ε, σε σχέση με τις ερωτήσεις και τα σχόλια που έγιναν ε, πρόκειται για μια πολύ ρεαλιστική έκθεση όπου θα ήθελα να απαντήσω με συγκεκριμένα και εστιασμένα σχόλια για τις ενέργειες της Κομισιόν σε αυτό το τομέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απόλυτα προσιλωμένη στην πρόθεση των ε, αλυσίδων ε, των υπεύθυνων αλυσίδων αξίας και όλοι εδώ προχωρούμε με διάφορες εσωτερικές και ε, με διάφορες ε, τρόπους ε, εσωτερικά και εξωτερικά της Ένωσης. Έχουμε πρόσφατα προτείνει νομοθεσίες που εστιάζουν σε περιβαλλοντικές και κοινωνικές θέσεις όπως ε, η οδηγία περί αποκάλυψης πληροφοριών από πλευράς των επιχειρήσεων για πολιτικές τους που αφορούν κινδύνους ε, για το περιβάλλον ή για θέματα κοινωνικά ή ε, θέματα των εργαζομένων ακόμα και για θέματα κατά της διαφθοράς. Η πρώτη σχετική έκθεση προβλέπεται για το 2018 και υπάρχουν και ρήτρες αναθεώρησης μέσα σε αυτή την οδηγία. Τώρα, όσον αφορά προγράμματα όπως το, το, το Ταμείο Vision Zero, το καταπίστευμα Ευρωπαϊκή Ένωση Ασία, έχουμε και εκεί προχωρήσει για σχετικά προγράμματα στην Ασία. Έχουμε ξεκινήσει δε διάλογο με τις χώρες παραγωγής ώστε να, να πιέσουμε τις δημόσιες αρχές να εφαρμόσουν τις διεθνείς συμβάσεις για τα εργατικά δικαιώματα και την προστασία του περιβάλλοντος μέσω διάβλων όπως πολιτική συζήτηση και την ρύθμιση ε, συν. Σε σχέση, έχουμε διάφορες εμπορικές δε πρωτοβουλίες ε, που ε, έχουμε δεσμευθεί για ευρωπαϊκές εμπορικές συμφωνίες. Στηρίζουμε την εργασία του ΣΑ και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και βεβαίως το σύμφωνο του Μπαγκλαντές. Καθώς προχωρούμε και προσπαθούμε να ενισχύσουμε τις δράσεις μας σε αυτές τους τομείς, θέλουμε να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις που ξέρουν πώς να στηρίξουν τη βιωσιμότητα στις στρατηγικές τους και να δημιουργήσουμε ε, να, μάλλον να βρούμε λύσεις αναπερίπτωση ε, προσπαθούμε να καλύπτουμε την βιωσιμότητα περισσότερο ως νοοτροπία και να στηρίξουμε για αυτά τα θέματα, καθώς και να χρησιμοποιήσουμε την ευρωπαϊκή μόχλευση σε μεγάλες εξαγωγικές χώρες. δεν θέλουμε να πάρουμε πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν στον αποκλεισμό χωρών που ε, παρουσιάζουν κίνδυνο βιωσιμότητας, αλλά που βασίζονται στο εμπόριο με την Ένωση και τις επενδύσεις από την Ένωση για να μπορέσουν να ε, προοδεύσουν. Έχουμε επενδύσει σημαντικά σε όλα αυτά και τώρα πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Χέντερσον. Κυρία Αρένα, θα θέλατε να ξαναπάρετε το λόγο. No, thank you. No. Όχι, ευχαριστώ. Ωραία, τέλεια. Ευχαριστώ την εισηγήτρια, ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μπορούμε να προχωρήσουμε κατευθείαν στο σημείο υπαριθμών 6 της ημερησίας διάταξης προκλήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά την εφαρμογή του ελεύθερου εμπορίου. Ο κύριος Κρίστοφερ Στίβεν, από το Overseas Development Institute θα μας παρουσιάσει μια μελέτη σχετικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων των αναπτυσσόμενων χωρών στον τομέα αυτό. Ε, κύριε Στίβεν, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ στην Επιτροπή μας από την Ισπανία. Διαδικαστικό, κυρία Πρόεδρε. Έχω ένα διαδικαστικό. Θα ήθελα να πω το εξής. Η συζήτηση για το σημείο 5 αναβλήθηκε επειδή περιμέναμε τον συνεισηγητή. Ε, παρεμβάλαμε το σημείο 4 αλλά επρόκειτο να επιστρέψουμε. Νομίζω λοιπόν ότι τώρα που ολοκληρώσαμε το σημείο 4 ε, θα πρέπει να πάμε στο σημείο 5 πάλι, όχι? Ναι, αλλά όπως βλέπετε ο κύριος Σιλικιώτης ακόμα δεν έχει καταφτάσει. Θα περιμένουμε λοιπόν και θα συζητήσουμε στο μεταξύ το σημείο 6. Α, μόλις κατέφτασε. Καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο να προεδρεύει κανείς υπό τέτοιες συνθήκες. Ζήτω συγγνώμη. Γεια σας κύριε Σιλικιώτη. Yes, I can fully understand. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Ο κύριος Σιλικιώτης, ε, καταλαβαίνετε, Προεδρεύω την αντιπροσωπεία με την Παλαιστίνη και έπρεπε να ολοκληρώσω και τις εργασίες για να καταφτάσω εδώ. Πρόεδρος, ε, ναι, Πηγαίνουμε από το ένα θέμα της ημερήσιας διάταξης στο άλλο. Σίγουρα δεν είναι βαρετή η συνεδρίαση η σημερινή. Λοιπόν... Μπορούμε λοιπόν να επανέλθουμε στο σημείο 5 της ημερησίας διάταξης. Κύριε Σιλικιώτη, Μόλις ακούσαμε παρουσίαση του συνεισηγητή σας, ε, του κυρίου Κοπουλάντε. Θα ήθελα τώρα να δώσω σε εσά το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω ελληνικά, τη μητρική μου. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, καταρχήν θέλω να καθιστορήσω και εγώ με τη σειρά μου τους συναδέλφους από τις χώρες της Αφρικής, της Καραβαϊκής και του Ελληνικού, για άλλη μια φορά στις Βρυξέλλες, Ιδιαίτερα θέλω να καλωσορίσω τον συνεισηγητή της έκθεσης μας για τη βελτίωση της αναπτυξιακής βοήθειας, τον κύριο Κοπουλάντε. Ε, είμαι, να σας πω στην ευχάριστη θέση, πως το προσχέδιο της έκθεσης μας σύζεται σε πολύ στερές βάσεις και η συνεργασία μας με τον κύριο Κοπουλάντε είναι πολύ παραγωγή. Στο κείμενο εντάχθηκαν αρκετές αναφορές που μας βρίσκουν απολύτως σύμφωνους για μας ε, οι ακόλουθε είναι ιδιαίτερα σημαντικέ. Η αρχή τη κυριαρχία των κρατών που λαμβάνουν αναπτυξιακή βοήθεια, δηλαδή οι χώρε που λαμβάνουν αναπτυξιακή βοήθεια να καθορίζουν τι αναπτυξιακέ προτεραιότητε και το μοντέλο για να τι εκτελέσουν. Συχνά αναπτυξιακά προγράμματα αποφασίζονται και σχεδιάζονται ανάλογα με τι προτεραιότητε των δωρητών χωρών. Συνεπώς, τα μοντέλα που εφαρμόζονται βασίζονται σε προηγούμενα επιτυχημένα προγράμματα τη χώρα ζωρετή, χωρί να δίνεται μεγάλη προσοχή στι τοπικέ ανάγκε και προτεραιότητε ή στο πλαίσιο το οποίο χρειάζεται να φέρουν αποτελέσματα. Το δεύτερο είναι η ανάγκη να διασφαλίζεται η κυριαρχία στο νερό και στην τροφή στι χώρε λήπτε τη αναπτυξιακή βοήθεια, όπω επίση και η ανάπτυξη των τομείων τη εκπαίδευση και τη υγεία σε δημόσιε υπηρεσίε. Το τρίτο είναι η προσήλεση στην αύξηση του προβλησμού που κάθε κράτος προσφέρει ως αναπτυξιακή βοήθεια στο 0,7 του ΑΕΠ του, μέσα στα πλαίσια των αναθεωρημένων στόχων της χιλιετίας. Σήμερα, η γενική παροχή αναπτυξιακής βοήθειας από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάνει στο 0,47% του ΑΕΠ. Το γεγονός πως η πάροχη βοήθεια δεν έφτασαν το 0,7% του ΑΕΠ του πριν το 2015 είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν 2-3 εκατομμύρια δολάρια για πρόθεση των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Γι' αυτό τον λόγο τα κράτη-μέλη της Ένωσης χρειάζεται να θέσουν σαφή χρονοδιαγράμματα για να πετύχουν το στόχο του 0,7 μαζί και το καθένα ξεχωριστά πριν από το 2030 αφού είναι ξεκάθαρο πως για επίτευξη των νέων αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας χρειάζονται επιπλέον μέσα. Το τέταρτο είναι η αναφορά για καταπολέμηση της στόχιας. Η μείωση της στόχιας είναι ένας από τους κύριους στόχους της αναπτυξιακής βοήθειας. Η μείωση της στόχιας είναι ένας από τους κύριους στόχους ε, που πρέπει να θέσουμε. Από το 2000 η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε το μεγαλύτερο μέρος του αναπτυξιακού της ταμείου σε εκείνες τις χώρες της, του ACP που το είχαν περισσότερο ανάγκη και ειδικότερα στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Αυτή τη στιγμή οι λιγότερο ανεπτυγμένε χώρε λαμβάνουν αυξημένο ποσοστό βοήθεια από 75,3% στο 1ο πακέτο του Ταμείου μέχρι το 81,1% του Ταμείου στο 11ο πακέτο. Την ίδια ώρα μειώθηκαν αυτά κονδύλια στις χώρες μεσαίου εισοδήματο από 5,5% σε 1,9% αντίστοιχα. Πέπτο, ιδιαίτερη σημασία έχει για μα η αναφορά για παροχή τη βοήθεια στα κράτη λήπτε ω χοργία και όχι ω δάνειο που να αυξάνει το εθνικό χρέο των χωρών του ACP. Πολιτικέ οικονομική χειραγώγηση των κρατών δεν εφόλεσαν πουθενά και τα παραδείγματα είναι πολλά τόσο εντό όσο και εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτό το φαινόμενο το έχουμε και στην ε, ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, δυστυχώ με τι πολιτικέ λιτότητα και μνημονίων που επιβλήθηκα στι χώρε τη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια, κυρίω του Ευρωπαϊκού Νότου, κατάφεραν ακριβώ το οικονομικό, τον οικονομικό νέο απικισμό, φτωχοποιώντα λαού και εργαζόμενου. Έβδομον, επίση κάτι που αποσχολεί ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2010 και μετά, είναι η μεταναστευτική πολιτική και ροή προσφύγων προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι με μεγάλη μας ικανοποίηση που βλέπουμε στο κείμενο την καταδίκη συμφωνιών μετανάστευσης. Της χρηματοδότησης δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στρατόπεδο συγκέντρωσης μεταναστών, γιατί μόνο έτσι μπορώ να τα χαρακτηρίσω, και προσφύγων σε χώρε κλειδιά στο πλαίσιο συμφωνία για αναπτυξιακή βοήθεια. Ω πολιτική ομάδα, εμεί είχαμε καταδικάσει και την παρόμοια συμφωνία που έγινε μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Τουρκία. Τέλος, βλέπουμε πολύ θετικά την αφορά για ανάγκη δεσμευτικών αρχών αναπτυξιακής βοήθειας στα πλαίσια του ΟΗΕ. Αυτές τις δεσμευτικές αρχές θα πρέπει να τις ακολουθούν τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές εταιρείε ή ιδιώτες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναβάλουμε την ετοιμότητα μας για μια παραγωγή συζήτηση και συνεργασία. Θα αντιμετωπίσουμε με παραγωγικό πνεύμα και επικοινωνικό πνεύμα όλες τις τροπολογίες που θα κατατεθούν και προσβλέπουμε επίση τη συζήτηση των τροπολογιών αυτών τόσο με τον συνάδελφο τον κύριο Κουμπουλάντη, όσο και με του άλλου συναδέλφου εδώ στην κοινωνιστική συνέλευση ίση εκπροσώπηση ΑΚΕ Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σιλικιώτη. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Ζήτω συγγνώμη που καθυστερήσαμε να καταφτάσουμε. Είχαμε τις μέρες ε, για την αναπτυξιακή βοήθεια και μιλούσαμε για την ε, αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας. Χαίρομαι που βλέπω στην έκθεση να γίνεται έκκληση για καλύτερο συντονισμό και για μεγαλύτερη οικειοποίηση από πλευράς των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να επιδιώξει τους στόχους αυτούς, ε, καθώς και όσον αφορά την ε, αρχή της αποτελεσματικότητας που αναφέρεται στην ε, Συμφωνία Ποσάν. Και θα πρέπει να τονίσουμε την λογοδοσία, το να εστιάζουμε στα αποτελέσματα και το να αναπτυχθούν συνεργασίες. Όπως γνωρίζετε, τον Νοέμβριο πραγματοποιήθηκε διάσκεψη υψηλού επίπεδου και πριν από τη συνάντηση αυτήν, Έγινε εκτενή συζήτηση του, ε, ε, της διακήρυξης ε, της συνάντησης αυτής και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Το θεματολόγιο για την βιώσιμη ανάπτυξη και οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αναφέρεται, αποτελούν ολοκληρωμένο όραμα με στόχο να εξαλειφθούν οι ανισότητες και γίνεται αναφορά στο θεματολόγιο της Αντίς απέπα, το πρόγραμμα δράσης της Αντίς Απέμπα, που έχει αλλάξει το τοπίο της ε, αναπτυξιακής βοήθειας. Ε, δεν είναι αλήθεια ότι η αναπτυξιακή βοήθεια είναι ο μόνος τρόπος να πετύχουμε τους στόχους ε, ανάπτυξης της χιλιετίας. Επίσης, στα συμπεράσματα της χιλιετίας, συγγνώμη, στα συμπεράσματα ε, του Συμβουλίου, ε, αναφέρεται ότι τα κράτη-μέλη έχουν ε, δεσμευτεί να πετύχουν τον στόχο, μέχρι, τον στόχο του ODA μέχρι το 2030. και έχουμε ανάπτυξη, σε, έχουμε αύξηση σε ονομαστικές τιμές όσον αφορά την ε, αναπτυξιακή βοήθεια προς ε, τις χώρες αυτές. Κάποιες χώρες μάλιστα δίνουν παραπάνω από το 0,7%. Μία από τις βασικές αρχές είναι η οικειοποίηση από πλευράς ε, των χωρών. Αναφέρεται ο κατακαιρματισμός της αναπτυξιακής βοήθειας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα ήταν υπέρ του κοινού προγραμματισμού, κάτι που έχει γίνει επιτυχώς σε 56 χώρες, εκ των οποίων 25 ε, είναι χώρες ΑΚΕ. Από αυτές τις 25 χώρες, οι 12 ήδη έχουν κοινή στρατηγική, προοδεύουμε λοιπόν. Ωστόσο, συνεχίζει να υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τις κυβερνήσεις εταίρους μας. Θα πρέπει λοιπόν και αυτό να το λαμβάνουμε περισσότερο υπόψη στην διαδικασία αυτή. Όσον αφορά ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, ε, τους πόρους αυτούς τους συζητάμε πάντα με τις χώρες εταίρους ε, και τα σχετικά προγράμματα τα εκπονούμε από κοινού. Προσπαθούμε λοιπόν ε, να λαμβάνουμε υπόψη μας την έννοια της εταιρικής σχέσης. Ε, μέρος της οικειοποίησης από τα κράτη είναι και η χρήση των συστημάτων των χωρών αυτών. Υπάρχουν ε, όμως κανόνες επιλαξιμότητας που συνδέονται με τη διαφάνεια και την ε, εποπτεία του προϋπολογισμού των τοπικών κοινοβουλίων. Επίσης, είναι απαραίτητη η κινητοποίηση διαφόρων πόρων για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους ε, στόχους της χιλιετίας μέχρι το 2030. Επίσης, θα ήθελα να σας μιλήσω για την πρόοδο που έχουμε σημειώσει όσον αφορά το θέμα της διαφάνειας η Κομισιόν και τα περισσότερα κράτη-μέλη ε, στο σύστημα ΑΙΑΤΑ δημοσιεύουν στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς ε, εκπόνησης του προπολογισμού και για να υπάρχει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με τον τρόπο αυτόν. Επίσης, ε, αυτήν την στιγμή εργαζόμαστε πάνω στο εργαλείο αυτό για τη διαφάνεια για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες των χρηστών. Ε, μπορεί λοιπόν ε, να έρθουμε σε επαφή, σε επαφή μαζί σας στο μέλλον πάνω στο θέμα αυτό. So, thank Σας ευχαριστώ πολύ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να ρωτήσω τους ευρωβουλευτές εάν υπάρχουν παρατηρήσεις. Παρακαλώ. Κυρία Συμπρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους δύο συνεισηγητές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δουλειά που έχουν κάνει. Χθε στη συζήτηση ε, λάβαμε συναγερμό σχετικά με την ε, τριγωνική σχέση και Ευρωπαϊκή Ένωση-Κίνα. έχει να κάνει με την ε, πραγματικότητα, με την πραγματική κατάσταση στις ε, διάφορες περιφέρειες. Και στη συζήτηση αυτή δόθηκαν σημαντικές πληροφορίες που θα πρέπει να ε, μας καθοδηγήσουν στην διαδικασία για τη διαμόρφωση της πολιτικής μετά το 2030 για να είναι πιο ισχυρή η πολιτική μας, ιδιαίτερα στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης. Πρέπει να παραδεχτώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει και κάνει πολλά πράγματα σε πολλές από τις χώρες μας. Σε πολλές ε, δράσεις πραγματοποιούνται σε χώρες ΑΚΕ, αλλά το ερώτημα είναι ποια είναι τα αποτελέσματα. Τελικά, δηλαδή, ποια είναι η συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξή μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την ε, πολιτική ανάπτυξης. Έχουμε 48 λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες σε όλο τον κόσμο, εκ των οποίων 31 ε, είναι χώρες ΑΚΕ. Ακούτε τι σας λέω. 41 από τα 49 κράτη είναι ε, ε, λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Είναι λοιπόν ένα γεγονός ιδιαίτερα δυστάριστο ότι μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας το 52 τα 100 των ε, χωρών ΑΚΕ συνεχίζουν να είναι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ω αν να μην ε, συμβαίνει τίποτα. Αυτό αδιαμφισβήτητα αποδεικνύει ότι η σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΚΕ και η βοήθεια που παρασχέθηκε δεν ε, έδωσε τα αποτελέσματα που θέλαμε να πετύχουμε. Και πρέπει να είμαστε ειλικρινεί όσον αφορά το θέμα αυτό. Υπάρχει μια δεύτερη ομάδα χωρών ΑΚΕ που είναι χώρες μεσαίου εισοδήματος. Κάποιες από τις χώρες ΑΚΕ στον κατάλογο αυτό είναι η ε, ε, Αγία Λουκία, ο ε, Αγίος Βικέντιος, η Ναμίμπια και η δική μου χώρα Σουρινάμ. το Τρίνιντατ και το Τομπάγκο έχουν, βρίσκονται ακόμα πιο ψηλά. Αυτά τα στοιχεία βασίζονται σε στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας. Κυρία Πρόεδρε, Αν εξετάσουμε αυτήν την ε, ομάδα των πιο ανεπτυγμένων χωρών εντός της ΑΚΕ, διαπιστώνουμε ότι απλά παρηγορούμεθα με στατιστικές για τις οποίες γνωρίζουμε ότι δεν μας δίνουν τη συνολική εικόνα. Έτσι αυταπατώμεθα εσκεμμένα. Πολλές αναλύσεις και μελέτες εμπειρογνωμόνων έχουν δείξει ότι υψηλό ΑΕΠ και υψηλό ΑΕΠ κατά κεφαλήν ε, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι δεν υπάρχει φτώχεια. Για παράδειγμα, το 10% του πληθυσμού μπορεί να κατέχει το 90% του πλούτου, ενώ το 90% να μοιράζονται μεταξύ τους το 10%. Αν εξετάσετε τις πιο ανεπτυγμένες χώρες της ε, ΑΚΕ, με βάση τον δείκτη για την ε, ανθρώπινη ανάπτυξη, πάλι η εικόνα δεν είναι ιδιαίτερα επιδοφόρα. Νομίζω ότι πρέπει να καταλήξουμε ότι η αποτελεσματικότητα της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι χαμηλή. Η οικονομική βοήθεια που παρασχέθηκε δεν έχει αντιμετωπίσει την φτώχεια. Ε, σε κάποιες περιπτώσεις ε, έχει κάνει τις χώρες αυτές ακόμα πιο εξαρτημένες σε πολλού τομεί. Ε, θα πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό και να έχουμε μια πιο ισχυρή και πιο αποτελεσματική συνεργασία. Επικεντρωθούμε λοιπόν στην ε, ανάπτυξη των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΚΕ και να αφήσουμε την Κίνα έξω από το σκηνικό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Άλλα σχόλια, παρακαλώ. Παρακαλώ, κυρία Ρένα. Ευχαριστώ. Θέλω να αντιδράσω σε αυτά που ακούσαμε μόλις. Κανείς δεν πίστεψε ότι με λιγότερο από 0,7% του Ευρωπαϊκού ΕΠ ε, θα μπορούσαμε να λύσουμε τα προβλήματα της φτώχειας της οποιασδήποτε υπήρου. Οπότε, οι κατηγορίες ε, για την αναπτυξιακή βοήθεια που δεν αντιμετώπισε τη φτώχεια στην Αφρική, την Καραβική και τον Ειρηνικό ε, είναι ίσως κάτι που λέτε έτσι πολύ εύκολα. Εγώ νομίζω ότι σίγουρα πρέπει να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα της βοηθειάς μας για να δούμε κατά πόσο επιτυχάνει τους στόχους, αλλά να το καθαρίζουμε αυτό ανάλογα με το βαθμό φτώχειας των χωρών στις οποίες αναφερθήκατε, δεν νομίζω ότι είναι η σωστή ανάλυση. Αν πράγματι θέλουμε να κάνουμε ορθή ανάλυση, τότε θα πρέπει να μιλήσουμε για το πώς αξιολογούνται οι πόροι των ίδιων αυτών χωρών από αυτές τις ίδιες χώρες και πώς οι πόροι αυτοί κατανέμονται από αυτές τις χώρες τους δικούς τους. Και αυτή την ανάλυση πρέπει να την κάνουμε. Το να λέμε ότι οι χώρες αυτές παραμένουν σε φτώχεια επειδή δεν είναι αποτελεσματική η δικιά μας η βοήθεια, νομίζω ότι είναι ένα διανοητικό εγχείρημα που κάνετε το οποίο σίγουρα δεν θα βοηθήσει τους μηχανισμούς ε, αναπτυξιακής βοήθειας που έχουμε στη διάθεσή μας. Πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Είναι αποτελεσματικοί οι μηχανισμοί αυτοί για τους στόχους μας. Αν δεν είναι, να τους βελτιώσουμε. Αλλά ας σταματήσουμε να λέμε ψέματα και να λέμε ότι φταίει το 0,7% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, γιατί αν ήταν 0,7% όντως αναπτυξιακή βοήθεια, τότε θα είχαν λυθεί και όλα τα προβλήματα που έχουν αυτές οι χώρες. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι αρχίζουμε να μιλάμε για σοβαρά πράγματα. Ο συνάδελφος εδώ δεν βάζει κανέναν στο ειδόλιο. Ο συνάδελφος προσπαθεί να παρουσιάσει την πραγματικότητα των πραγμάτων όσα έχουν σήμερα. Λιγότερο από 0,7% θα μπορούσε να φτάνει. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι συγκρίνουμε με άλλες εταιρικές σχέσεις που έχουμε. Τι θα έπρεπε να έχουμε στη διάθεσή μας από την ευρωπαϊκή βοήθεια. Το έχουμε? δεν μπορούμε να δεχτούμε η εκτέλεση, η παρακολούθηση της ευρωπαϊκής βοήθειας στις χώρες ΑΚΕ να είναι αποτυχία. Δεν πρόκειται για την ποσότητα, πρόκειται για τη χρήση της ποσότητας των χρημάτων. Αναφέρθηκε στην, στην Κίνα. Γιατί όσον αφορά τις χώρες ΑΚΕ, η Κίνα είναι μια πραγματικότητα είναι μια συγκεκριμένη πραγματικότητα, απτή, που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των χωρών ΑΚΕ και του πληθυσμού των χωρών ΑΚΕ. Ενώ η ευρωπαϊκή βοήθεια για τις χώρες ΑΚΕ παίζεται στην Ευρώπη και τους ε, κυβερνώντες, βέβαια με τις πολυεθνικές και τα λόμπι, με αποτέλεσμα οι πληθυσμοί των χωρών ΑΚΕ να μην υποφελούνται από αυτή τη βοήθεια. Και αυτό είναι που λέμε σήμερα, ότι μαζί εμείς και εσείς πρέπει να επανακαθορίσουμε τον τρόπο χρήσης της βοήθειας αυτής. Αυτό θέλουμε. Και σας εγγυώμαι ότι το 0,7% είναι και παρά αρκετό. Πάνω από 42 χρόνια έχουμε εταιρική σχέση. Τα προβλήματα όμως παραμένουν. Και πρέπει να αναρωτηθούμε όντως γιατί. Θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε τι συμβαίνει. Και το λέω ότι αν συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο κι άλλο, τότε Ας αφήσουμε τους Ευρωπαίους, έχουν προβλήματα. Το Παρίσι είναι δύσκολο να έχει κανείς 5.000 στο Σαντενί. Όμως, πρέπει να δούμε ποιος διαχειρίζεται τα χρήματα. Εγώ θα προτιμούσα τη βοήθεια αυτή να τη δώσετε σε κάποιον στο Σαντενί, αν αυτό τη χρησιμοποιήσει καλύτερα και μπορέσει να υποφεληθεί, παρά να πηγαίνει σε εμά. Αυτό είχα να πω. Τίποτα άλλο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε και μετά ποιος τώρα η Γουινέα και μετά η Νότια Αφρική. Εντάξει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η συζήτηση είναι ιδιαίτερα καρποφόρα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της βοήθειας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι η πιο αποτελεσματική βοήθεια είναι αυτή που μας βοηθάει να μην χρειαζόμαστε βοήθεια. Και την βοήθεια έτσι όπως την γνωρίζουμε σήμερα δεν είναι μια βοήθεια που μας βοηθάει να μην τη χρειαζόμαστε πια. Και θυμάμαι ότι το Σεπτέμβριο του 1978 στην πρώτη διάσκεψη του ΕΣΤΟ Παρίσι για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, που τότε ήταν 29 στον κόσμο, τότε ήταν που αποφασίσαμε για το 0,7% του ΑΕΠ των αναπτυγμένων χωρών για να αντιμετωπιστεί η φτώχεια ανά τον κόσμο. Σήμερα είμαστε 48 οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Να, ο δείκτης της αποτελεσματικότητας της ευρωπαϊκής βοήθειας οι χώρες μας γίνανε χώρες οι οποίες ε, παρέχουν πρώτες ύλες. Η μάχη που δίνουν οι χώρες αυτές είναι τεράστια για να μπορούν να έχουν κάποια προστιθέμενη αξία οι Και όπως το είπε η κυρία Μαρία Ρενά, η συζήτηση έχει να κάνει με την τοπική μεταποίηση των χωρών. Δηλαδή, καμία πρώτη ύλη δεν είναι αποτελεσματική αν δεν έχει προηγουμένως μεταπηθεί. Είτε πρόκειται για το βοξίτη, είτε πρόκειται για οτιδήποτε άλλο. Η χώρα μου εξάγει πολύ βοξίτη. Όσο συνεχίζουμε 26 δολάρια να πουλάμε τον τόνο βοξίτη, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε ένα κιλό αλουμίνιο που να εξάγεται από τη χώρα μας, με πολύ καλύτερη τιμή, ε, δεν θα βγούμε από αυτή την κατάσταση. Άρα λοιπόν υπάρχει η βούληση, φαίνεται, οι χώρες που δίνουν την πρώτη ύλη να παραμείνουν. Να μην μπορέσουν να μεταπίσουν. Δεν μπορούμε να μεταπίσουμε εμείς την πρώτη ύλη. Δείτε τι γίνεται με τον καφέ. Η χώρα που εξάγει περισσότερους σπόρους καφέ, εισάγει τον καβουρδισμένο καφέ για να το χρησιμοποιήσει. Ε, λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι η καλύτερη βοήθεια είναι εκείνη η οποία θα μας βοηθήσει να μην χρειαζόμαστε πια βοήθεια, που θα μας βοηθήσει να μπορούμε εμείς τις πρώτες ύλε που διαθέτουμε να τις μεταποιούμε και να μπορούμε να τις εξάγουμε σαν κάτι άλλο. Ευχαριστούμε. Η Νότια Αφρική τώρα. Ευχαριστώ πολύ, αξιότιμη Πρόεδρος. Επιτρέψτε μου να επωφεληθώ από την ευκαιρία αυτή για να συμμετάσχω και εγώ στη συζήτηση. Ευχαριστούμε για την έκθεση που παρουσιάστηκε από τους δύο εισηγητές. Έχω να πω το εξής. Θέλω να θίξω ένα ζήτημα Δεν είναι δυνατόν να ερχόμαστε εδώ και να λέμε ψέματα για την κατάσταση. Νομίζω ότι συμφωνούν οι συνάδελφοι. Δεν είναι δυνατόν να ερχόμαστε από τόσο μακριά εδώ στις Βρυξέλλες και να λέμε ψέματα ότι τα 42 χρόνια εταιρική σχέση δεν έχει βοηθήσει τους λαούς μας. οποιαδήποτε εταιρική σχέση πρέπει να είναι ισότιμη. Είτε διαθέτεται πόρους, είτε δεν διαθέτεται πόρους. Αν είναι μια πραγματική εταιρική σχέση, τότε είναι μια εταιρική σχέση που θα διασφαλίζει ότι και οι δύο πλευρές είναι ισότιμες. Ότι και αυτοί οι οποίοι παίρνουν την βοήθεια αντιμετωπίζονται ισότιμα. Και θα δώσω ένα παράδειγμα που είπε και ο συνάδελφος από τη Γουινέα. Στις χώρες μας, οι φυσικοί πόροι μας εξορίσονται και φεύγουν από τις χώρες μας και έρχονται σε εσά. Αν λοιπόν πρόκειται για μια πραγματική εταιρική σχέση, αυτές οι χώρες ΑΚΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να μεταποιούν, να επεξεργάζονται τους ε, πόρους τους, τις πρώτες ύλε τους τόπου. Αλλιώς δεν πρόκειται για πραγματική εταιρική σχέση. Και δεν μπορεί να λέτε ότι λέμε ψέματα όταν εξακολουθούν υπάρχουν τόσοι άνθρωποι στις χώρες μας οι οποίοι υποφέρουν από πείνα, από ασθένειες. Δεν μπορεί να εξαρτώμαστε Ισαΐ οι χώρες της Αφρικής, Καραϊβικής, ε, Ειρηνικού από τη βοήθειά σας. Χρειαζόμαστε μια εταιρική σχέση και μια βοήθεια η οποία να μας βοηθάει με προγράμματα στις χώρες μας. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι γι' αυτό. Προγράμματα τα οποία δεν έχουν τελικά θετικές επιπτώσεις στις χώρες μας, βεβαίως και δεν μας βοηθούν και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Πρέπει, συνεπώς, να αποκτήσουμε τα κατάλληλα προσόντα της δεξιοτεχνίες εκείνες που θα μας βοηθήσουν να εκμεταλλευόμαστε σωστά και να επεξεργαζόμαστε τους πόρους μας. Με εκπαίδευση, με κατάρτιση. Είναι η συλλογική μας ε, θέση αυτή των χωρών και ότι οποιαδήποτε βοήθεια πρέπει να έχει και ένα στοιχείο ισοτιμίας. Οποιαδήποτε χώρα δικαιούχος πρέπει να εκτιμάει και εκείνη, να αξιολογεί και εκείνη το πρόγραμμα εκείνο το οποίο υλοποιείται στην συγκεκριμένη χώρα. Δεν είμαστε έτσι διακοσμητικά στοιχεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή για οποιονδήποτε άλλον. Ευχαριστώ. Το Μπουρούντι τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κι εγώ θέλω να αναφερθώ για στην αποτελεσματικότητα της βοήθειας. Ο αριθμός των δικαιούχων στις χώρες ΣΑΚΕ είναι τέτοιος που δείχνει ποια είναι η ανάγκη. Το 0,7% μάλλον το 0,47% πρέπει να αυξηθεί αν θέλουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες. Έπειτα, όχι μόνο δεν φτάνει, αλλά επιπλέον χρησιμοποιείται και σε τομείς που δεν έχουν επιλεχθεί σωστά. Μάλλον γιατί δεν έχουν ερωτηθεί επαρκώς οι δικαιούχοι. Η βοήθεια λοιπόν θα πρέπει να δίνεται στις πιο φτωχές χώρες ώστε αυτές να περάσουν από το καθεστώς της φτωχής χώρας σε εκείνο της αναδυόμενης χώρας. Το είπαν και οι συνάδελφοι ότι δυστυχώς έχουν αυξηθεί οι χώρες στην κατηγορία των φτωχών χωρών. Θα σας δώσω το παράδειγμα της δικιάς μου χώρας, του Μπουρούντι. Έχουμε πάρα πολύ νίκελ εμείς, το οποίο βρίσκεται εκεί, αλλά δεν μπορούμε να το επεξεργαστούμε, γιατί δεν διαθέτουμε ενέργεια. Οπότε δεν θα πρέπει η ευρωπαϊκή βοήθεια να προσανατολιστεί έτσι ώστε να δημιουργηθούν υποδομές που να μας επιτρέπουν να έχουμε αρκετή ενέργεια για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε όλες αυτές τις ποσότητες νίκελ που διαθέτει το επεδαφός μας. Θέλω να πω ότι η επιλογή, ο προσανατολισμός της βοήθειας θα έπρεπε να κατευθυνθεί αλλού σε προγράμματα τα οποία να βοηθήσουν τις στοχές χώρες να περάσουν στο στάδιο των αναδιόμενων χωρών. Αυτό είχα να πω. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Το πράσινο κροτήρι. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ε, θέλω και εγώ να συμβάλλω σε αυτή τη συζήτηση για την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών ΑΚΕ σε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα που είναι η καταπολέμηση της στόχιας. Πιστεύω ότι στη διάρκεια των ετών έχουμε υιοθετήσει ένα πρότυπο το οποίο έχει αναπαράξει τις τα ίδια αποτελέσματα και Αυτό γιατί έχει χρησιμοποιηθεί το ίδιο πρότυπο ανάπτυξης και βοήθειας. Και χρόνο με το χρόνο η κατάσταση της φτώχειας παραμένει ίδια. Και εδώ πρέπει να πω ότι η φτώχεια δεν θα πρέπει να τη διαχειριστούμε πλέον, αλλά να την εξαλείψουμε. Και για να την εξαλείψουμε πρέπει να ανακαθορίσουμε τον τρόπο, το πρότυπο, το αναπτυξιακό που χρησιμοποιούμε. Και επίσης οι ενισχύσεις που λάβαμε ε, θα, θα πρέπει διαφορετικά να χρησιμοποιηθούν για αυτούς τους στόχους. Ε, θα πρέπει να εστιάσουμε στην παιδεία και κυρίως στη δημιουργία ενός οικονομικού περιβάλλοντος, ενός εμπορικού περιβάλλοντος που να είναι σε θέση να δημιουργήσει και να, καλέσει, να προσελκύσει μάλλον περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις ώστε να μπορούμε να έχουμε περισσότερη απασχόληση και ο κόσμος να έχει μεγαλύτερα έσοδα, εισοδήματα. Έτσι μπορούμε να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια και ήθελα λοιπόν ε, αυτά να πω. Στην ουσία αυτό που χρειάζεται είναι να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης και έτσι να μπορέσουν να αξιοποιηθούν και ε, τα, ε, να αξιοποιηθεί ο κόσμος. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να είμαστε συνεπείς με τους αυτούς μας. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι είναι ανεπαρκής η βοήθεια. Α πούμε ότι δεν χρησιμοποιείται καλά. Αν δεν χρησιμοποιείται καλά, τότε γιατί να την αυξήσουμε, αν δεν χρησιμοποιείται καλά. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, η ερώτηση που πρέπει να κάνουμε είναι τι ανάπτυξη θέλουν πραγματικά οι χώρες ΑΚΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν νομίζω ότι επέβαλε κανένα μοντέλο ανάπτυξης. Εσείς πρέπει να κάνετε προτάσεις και βάσει των προτάσεων αυτών θα εξετάσουμε τελικά ορθά τα πράγματα. Συνεπώς, τι προτάσεις έχετε εσείς να κάνετε προκειμένου η βοήθεια που δίνεται στις χώρες ΑΚΕ να είναι αποτελεσματική, να χρησιμοποιείται ικανοποιητικά υπέρ του πληθυσμού στον οποίο αναφέρεστε. Έτσι πρέπει να θέσουμε το ζήτημα. Να μην λέμε ότι δεν είναι αρκετή βοήθεια, ότι θέλουμε παραπάνω βοήθεια, μετά να λέμε ότι δεν χρησιμοποιείται καλά, ότι υπάρχει σπατάλη, ότι οι κυβερνήσει ε, χρησιμοποιούν τα χρήματα αυτά σε βάρο του πληθυσμού. Δεν πρέπει να λέμε αυτά. Πρέπει να κάνουμε προτάσει. Γιατί εδώ δεν είμαστε στο στάδιο που θα λέμε μόνο τι δεν πάει καλά. Πρέπει να λέμε και τι προτείνουμε για να πάει καλά ή για να πάει καλύτερα. Αυτό είχα να πω εγώ. Παρακαλώ. Εσείς δεν καταφέρνω να διαβάσω το όνομά σας, αλλά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πώς θα είναι αποτελεσματική η βοήθεια για τις αφρικανικές χώρες, τις χώρες ΑΚΕ κυρίως. Εδώ θέλω να πω πώς πρέπει να προσανατολιστεί η βοήθεια αυτή και να κάνω και μια διάγνωση για κάθε χώρα, για κάθε περιοχή πιο σωστά. Στις χώρες ΑΚΕ, λοιπόν, γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα εκπαίδευσης, υγείας και σε άλλες βασικές υποδομές. Νερό, ηλεκτρισμός και δρόμοι. Προκειμένου λοιπόν η βοήθεια να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει οι ευρωπαϊκές χώρες πριν δώσουν χρήματα για βοήθεια, διακόπτει τον ομιλητή κάποιος. Έλεγα λοιπόν ότι στις χώρες ΑΚΕ χρειάζονται βασικές υποδομές. Αλλού υπάρχουν αυτές οι βοήθειες. Αν λοιπόν την ευρωπαϊκή βοήθεια τη στρέψουμε προς τις αφρικανικές χώρες, χώρες ΑΚΕ, προς τις υποδομές που δεν έχουν, εκεί θα βοηθήσει η βοήθεια. Αν όμως δεν κάνουμε τη διάγνωση για το ποιες είναι οι ανάγκες της κάθε χώρας, της κάθε περιοχής, πριν δώσουμε τη βοήθεια, μπορεί να κάνουμε λάθος. Μερικές φορές οι χώρες διαθέτουν ήδη κάτι. Κάποιες έχουν πολύ αδύναμους πόρους, που σημαίνει ότι αν η βοήθεια δεν προσανατολιστεί σωστά, οι θετικές επιπτώσεις της βοήθειας στην οικονομία και την κοινωνική υποδομή της χώρας θα χαθεί. Άλλος κανείς. Παρακαλώ. Εσείς. Καλησπέρα σας. Από τη Γουινέα Μπισάου. Αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι θα μπορούσαμε να διαμορφώσουμε διαφορετικά τη συζήτησή μας και να την προσανατολίσουμε και διαφορετικά. Διότι Όντως έχουμε λάβει τις ενισχύσεις, τη βοήθεια, αλλά στην πραγματικότητα η ανάπτυξη της κάθε χώρας είναι ευθύνη και αρμοδιότητα της κυβέρνησης της. Η βοήθεια είναι συμπληρωματική, κατά τη γνώμη μου. Εγώ, ίσως επειδή προέρχομαι από μια χώρα με χρόνια αστάθεια, τελείως χρόνια αστάθεια, διαπίστωσα πως δυστυχώς δεν μπορούμε να αποσυνδέσουμε την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, την καταπολέμηση της στόχιας από την πολιτική. Ορισμένες χώρες όπως, που, έχουν μάλλον το ίδια μοντέλα οικονομικής βοήθειας κατάφεραν να βγουν από την κατηγορία των αδύναμων και υπανάπτυκων χωρών και να ε, μετατραπούν σε χώρες μιας μέσης ανάπτυξης. Αν αναλύαμε την κατάσταση θα, θα καταλήγαμε στο συμπέρασμα ότι όντως με παράδειγμα την Γουινέα Κόνακρη, ε, όπου εμείς συνεργαζόμαστε γιατί την, ε, εκεί κάνουμε τη μεταποίηση τη, των πρώτων μας υλών, ε, θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε καλύτερα. Όμως πρέπει να κάνουμε και την εξή ανάλυση. Οι χώρες που κατάφεραν να αναπτυχθούν είναι χώρες οι οποίες είναι προσιλωμένες στην καταπολέμηση της διαφθοράς, είναι χώρες που είναι προσιλωμένες στη καλή χρηστή διαχείριση και προσιλωμένες στη δημοκρατία. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλέσω να αναλύσουμε και αυτή, αυτό το χαρακτηριστικό για να μπορέσουμε οι ίδιοι να μιλήσουμε για τις ευθύνες των ίδιων μας χωρών. Θα πρέπει λοιπόν να προσιλωθούμε στις δημοκρατικές αξίες, στις αξίες της καταπολέμησης της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής, της φοροαπάτης, να προσιλωθούμε στην καταπολέμηση της στόχιας, και κατά, εν πάση περιπτώσει, όλων όσων ε, συμβάλλουν στον πλουτισμό ορισμένων και στη φτώχυνση των πολλών. Εντάξει οικονομικέ οικονομικές αναλύσεις, αλλά να συνδέσουμε τη συγκεκριμένη πολιτική ε, ε, κρίση με το θέμα της φτώχειας της χώρα μας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να σχολιάσει τα όσα είπαν οι τα μέλη της ε, συνέλευσης, η Κομισιόν. Ακούστε, το θέμα εδώ νομίζω είναι η δημοκρατική και συμπεριληπτική οικειοποίηση. Το είπα και πριν. Εμείς ε, θέλουμε τη δημοσιονομική στήριξη. Για να υπάρχει δημοσιονομική στήριξη ε, πρέπει να εκπληρώνονται κάποιες βασικές προϋποθέσεις που είναι οι δημοκρατικές αξίες. Το προείπα. Για το προγραμματισμό ε, των κοντιλίων του ΕΤΑ και εδώ μιλάω από την ιδιότητα μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν μιλάμε απλά για την απόφαση που θα πρέπει να ληφθεί που θα πάνε τα χρήματα. Είναι μια διαδικασία ε, όπου συμμετέχουν όλοι. Άρα και η κοινωνία των πολιτών, οι κυβερνήσεις, οι διάφοροι οργανισμοί και ε, κυβερνητικές ε, οργανώσεις, αλλά και το κοινοβούλιο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται Άρα, στην όλη συζήτηση για το πώς μπορούμε να μειώσουμε τη φτώχεια, η απάντηση είναι να είμαστε συμπεριληπτικοί, όλοι δηλαδή να συμμετέχουν και να έχουμε περισσότερη εταιρική σχέση. Η πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για τα σχόλιά τους, τις παρατηρήσεις τους. Θέλετε να δευτερολογήσετε, βεβαίως, ευχαρίστως. Ε, κύριε Σιλικιώτη, παρακαλώ. Very short, yeah. Uh, I will speak Greek. Uh, πρέπει να πω ότι ε, εγώ χαίρομαι γιατί κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Και να σας πω ότι προσυπογράφω σχεδόν τα περισσότερα που είπαν οι εκπρόσωποι από τη Σάκη και ο εκπρόσωπος από το Σουρινάμ και από τη Γουινέα και από το Μπουρούντι και από, το, από την Νότια Αφρική. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δεν φτάνει η βοήθεια. Είναι το μοντέλο, είναι το πρότυπο της βοήθειας. Και είναι σωστό αυτό που είπε ο εκπρόσωπος της ε, Ουινέας ότι ε, ε, δεν πρόκειται για την ποσότητα, είναι για τη χρήση της βοήθειας. Και όντως η βοήθεια πρέπει να δίνεται για να βοηθήσει τις χώρες να ξεφύγουν από τη φτώχεια. Είναι επίσης αλήθεια ότι ε, μπορεί σε κάποιες χώρες να μιλούμε για ανάπτυξη, αλλά την ίδια ώρα να, το ερώτημα πρέπει να βάζουμε ανάπτυξη για ποιου. Ποιο οπεφελείται από αυτήν την ανάπτυξη. Γιατί την ίδια ώρα διευρύνονται οι ανισότητε. Δηλαδή έχουμε το μοντέλο οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί να γίνονται φτωχότεροι. Και δεν λέμε πράγματα που υπάρχουν μόνο στη ΣΑΚΕ. Επειδή τη χάνει να προέρχομαι από τον νότο τη Ευρώπη, το ίδιο μοντέλο χρησιμοποιείται και για τον νότο τη Ευρώπη. Δίνεται βοήθεια, η οποία αντί βοήθεια να ε, βοηθά τι χώρε να ξεφεύγουν από την κρίση και την, ε, από την ύφεση, να οδηγούν το όλο ένα και περισσότερο στην κρίση και στην ύφεση, με ψηλά ποσοστά ανεργία, με διεύρυνση των ανισοτήτων, με σπρόξιμο μεγάλη μερίδα του πληθυσμού στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Άρα το ζητούμενο είναι να δούμε, ναι, ε, το, μπορεί να αυξηθεί η βοήθεια, αλλά το κυριότερο πρέπει να δούμε το μοντέλο που δίνεται αυτή η βοήθεια. Και κλείνω λέγοντας ότι ναι, μέσα μαζί με τον συνάδελφο Κουπουλάντε. Αυτό που προσπαθούμε μέσα από αυτή την έκθεση είναι να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας ώστε να αλλάξει αυτόν το πρότυπο, αυτόν το μοντέλο ε, της ε, οικονομικής βοήθειας και θεωρώ ότι βεβαίως με ε, μια έκθεση που είναι τόσο σύντομη δεν μπορεί να περιλάβει στα πάντα αλλά ακριβώς προσπαθούμε να συμβάλλουμε από τη δική μας πλευρά ώστε να υπάρξει μια οικονομική βοήθεια, ένα πρότυπο ε, βοήθειας ε, για να βοηθήσει στην ανάπτυξη των χωρών στο να ξεφύγουν ακριβώς αυτές οι χώρες από την υπανάπτυξη, τη φτώχεια και την εξαθλίωση των λαών τους. Ευχαριστώ Πρόεδρε για, την, ε, για που μου έδωσε τον λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σιλικιώτη. Κύριε Κοπουλάντε, παρακαλώ, έχετε το λόγο τώρα. Κύριε συμπρόεδροι, κυρίες συμπρόεδροι, αξιότιμοι συνάδελφοι, ήταν μια υψηλού επίπεδου και πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για ένα άκρο σημαντικό ζήτημα διότι είναι ένα ζήτημα το οποίο προσδιορίζει τον ιστό και την, τον λόγο ύπαρξης ε, των σχέσεών μας. Αυτό το θέμα, αγαπητές κυρίες συμπρόεδροι, καθορίζει και το μέλλον, το μέλλον της ανθρωπότητος. Διότι αν πράγματι η Ευρώπη πιστεύει ότι μπορεί να συνεχίσει να ζει πλήρη αυθονία αφήνοντας ε, τις υπόλοιπες ε, χώρες ε, να ζουν σε πλήρη φτώχεια δεν μπορείτε πάνω, να κάθεστε πάνω σε μια χωματερή και να πίνετε σαμπάνια όχι. Πρέπει να το κάνετε είτε στην πρώτη θέση του αεροπλάνου, είτε σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η προσέγγιση στην ανάπτυξη θα πρέπει να είναι μια προσπάθεια αναβάθμισης, διότι η αμοιβαία ευημερία είναι προς αμοιβαίο όφελος, προς όφελος όλων των εταίρων. Και πραγματικά με λύπησε αυτό που άκουσα. Να δω ποιος το είπε. Ο σύμβουλος ε, για το ε, διεθνές εμπόριο και τις παγκόσμιες ε, αλυσίδες αξίας και είπε ότι δεν είναι αλήθεια αυτά τα στοιχεία. Μα εμείς δεν λέμε ψέματα. Στοιχεία είναι αυτά. Ότι δεν εξετελέστησαν οι δεσμεύσει για το 0,7 της, ε, του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος. Δεν λέμε ψέματα. Είναι γεγονός αυτό. Το 0,7% του Ευρωπαϊκού, λέει ο μιλητή ακαθάριστου Δεν λέμε ότι θα λύσει το πρόβλημά μα 100%, ε, τα προβλήματά μα 100% σε καμία περίπτωση. Ούτε ε, πουθενά το έχουμε γράψει. Αντίθετα, στα ψηφίσματά μα λέμε ξεκάθαρα ότι οι ε, αποδέκτερε χώρε θα πρέπει να ορίσουν τι δικέ του αναπτυξιακέ προτεραιότητε τις δικέ τους αναπτυξιακές επιτακτικές ανάγκες και τις αντίστοιχε αναπτυξιακές στρατηγικές. Και αυτό το πράγμα το ξεκαθαρίσαμε και στην έκθεσή μας και στα ψηφίσματά μα το λέμε. Και σε αυτήν την έκθεση δίνουμε έμφαση στην ανάγκη για επενδύσει. Και λέμε ότι θα πρέπει να πάνε τα χρήματα στην δημιουργία υποδομών, στην παιδεία, στην υγεία, ώστε μακροπρόθεσμα οι χώρες ΑΚΕ να έχουν τις δικέ τους δυνατότητες και ικανότητες για να μπορεί η οικονομία τους να αυξηθεί και να καταπολεμηθεί φτώχεια. Από μέσα στην ίδια τη χώρα να γίνονται, από την ίδια χώρα να ξεκινούν οι προσπάθειες και στην πρώτη μου παρέμβαση το τόνισα και είπα ότι η βοήθεια θα πρέπει να βρει το δρόμο της και δεν θα πρέπει να μπει ε, στην ε, δεν θα πρέπει να διονυστεί, αλλά κάποια στιγμή να αντικατασταθεί από πιο μόνιμες εμπορικές συμφωνίες. Και θέλουμε εμπορικές σχέσεις δυνατότητες με τις χώρες ΑΚΕ, ώστε να μπορούμε να προσθέσουμε την αξία μας στις δικές μας πρώτες ύλες. Για να έχουμε περισσότερη αξία. αν ε, συνεχίσουμε να διατηρούμε αυτή τη σχέση ακριβώς ε, που ουσιαστικά είναι προμηθευτές πρώτων υλών οι χώρες ακές της βιομηχανής Ευρώπη, αυτό δεν είναι βιώσιμο ως πρακτική και πολιτική. Θα έρθει μια μέρα που θα, πάρουμε ε, που θα πάρουμε μια απόφαση εμείς προμηθευτές πρώτων υλών σε ό,τι αφορά τα οικονομικά μέσα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους πήραν το λόγο. Αλλά ήθελα να εκφράσω κάποιες ε, επιφυλάξεις για τη συλλογιστική. Πίσω από αυτό που λέμε κοινωνία των πολιτών. Η συμπρόεδροι θα γνωρίζετε ότι η κοινωνία των πολιτών, οι συνοργανώσει αυτέ, ε, στο μεγαλύτερο μέρο, για να μην πω εξ χρηματοδοτούνται από τι δωρήτερε χώρε. Ποια ατζέντα ε, προωθούν την ατζέντα αυτών των χωρών. Τελικά, ε, Γιάννης ε, κερνάει, Γιάννης πίνει. Αυτός που χορεύει, που υπαγορεύει τη μουσική χορεύει, ποιος θα καθορίσει την ατζέντα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που επιβάλλουν τι απόψει, επιβάλλονται στι διάφορε κοινωνίε και κάνουν ε, την απόπειρα να ε, και τείνουν να υποστηρίζουν δόγματα τα οποία μπορεί να είναι προς όφελος αυτών ε, που τους πληρώνει. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά. λέμε ότι οι χώρε για αποδέκτες θα πρέπει να μπορούν να ε, καθορίζουν τη δική τους ατζέντα. Ποιοι πήραν την εντολή από το λαό. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να καθορίζουν την ατζέντα για το λαό που τους έδωσε την εντολή. Κάποιες φορές ε, η κοινότητα πολιτών έχει την τάση να παραπλανά την προσοχή, να τη στρέφει σε άλλα θέματα, τα ήπια ζητήματα όπως τα λέω εγώ, σε σχέση με τα πολύ επίγοντα ζητήματα. Αυτό που θέλει η περιοχή μας είναι ανάπτυξη πραγματικής οικονομίας και εκεί πρέπει να πάει βοήθεια. Γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος να περάσει στη λύθη κάποια στιγμή και να ξεχαστεί και να σταματήσει αυτή η πολιτική. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας ε, θυμίσω ότι το ψήφισμα θα το ψηφίσουμε στην επόμενη Ολομέλεια στη Μάλτα τον Ιούνιο. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η Τετάρτη 10 Μαΐου στις 12 ε, το μεσημέρι. Προχωράμε στο σημείο 6 της ημερησίας διάταξης. Ο κύριος Στίβενς είναι εδώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ στην Επιτροπή μας. Η Επιτροπή Ανάπτυξης της ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησε την εκπόνηση μελέτης, όπου στόχο έχει να εξετάσει τις διπλές προκλήσεις των ατισόμενων χωρών ε, κατά την εφαρμογή των ε, συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου. Και θα Πρέπει να εξεταστεί η ανάγκη για, την, ε, για τον εξυγχρονισμό των ε, διοικήσεων ε, των φορολογικών αρχών για να μπορούν να επωφεληθούν από το πιο απελευθερωμένο εμπόριο. Η μελέτη αυτή αναμένεται να προτείνει τρόπους να ξεπεραστούν οι προκλήσεις αυτές και θα ε, ληφθεί υπόψη κατά τις ε, συζήτηση που, που πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή εντό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην ε, κοινή κοινοβουλευτική συνέλευση και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη από την αρχή το Κοινοβούλιο εξέφρασε ανησυχίες του σχετικά με το πιθανό αντίκτυπο των συμφωνιών και τις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές των χωρών εταίρων για κάποιες χώρες ΑΚΕ οι, φορολογικοί, οι ε, δασμοί, οι τελωνιακοί δασμοί αποτελούν ε, σημαντικό κομμάτι των ε, εσόδων τους και βραχυπρόθεσμα θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την απώλεια αυτών των εσόδων, διότι τα ωφέλη μάλλον θα αργήσουν να φανούν. Δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Στίβενς χωρίς καθυστέρηση για να μας παρουσιάσει τη μελέτη του. Uh, Κυρία Συμπρόεδρε, ε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, ε, ε, Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε την δυνατότητα να σας παρουσιάσω αυτήν την μελέτη. Όπως αναφέρθηκε στις εισαγωγικές παρατηρήσεις της Συμπροέδρου, η μελέτη έχει κυρίως να κάνει με τις επιπτώσεις στα έσοδα της απελευθέρωσης του εμπορίου, ε, αρχικά στα πλαίσια των ε, συμφωνιών αυτών, αλλά γενικά στο πλαίσιο των ε, εμπορικών συμφωνιών που συνυπογράφουν οι χώρες ΑΚΕ. Το θέμα λοιπόν είναι πώς μπορεί να μεταβληθεί η φορολογική βάση τη στιγμή που προοδεύουμε στα ζητήματα αυτά. Η μελέτη βασίζεται σε εξέταση πάνω από 70 μελετών σχετικά με τις επιπτώσεις στα έσοδα των συμφωνιών εταιρικής σχέσης. Έχουμε πάρει λοιπόν στοιχεία από αυτές τις μεταμελέτες. Πολύ σημαντικό ε, θέμα στο οποίο θα επανέλθω αργότερα είναι ότι όλα τα στοιχεία αυτά αποτελούν προβλέψεις. Δεν ε, αποτελούν ε, εξέταση των όσων έχουν ήδη συμβεί, κυρίως επειδή δεν έχει συμβεί τίποτα ακόμα. Ούτε βασίζονται τα στοιχεία αυτά σε ιδιαίτερα στεναρή βάση δεδομένων σε χώρες που έχουν απελευθερώσει το εμπόριο. Οι προβλέψεις δεν είναι κακές, ε, οι προβλέψεις είναι δεν είναι κακό πράγμα, είναι σημαντικό πράγμα. Αλλά εάν στις αρχές του έτους έχει γίνει πρόβλεψη ότι η ανάπτυξη στη χώρα σας ε, θα είναι του ύψους 1-2% και στο τέλος ε, της χρονιάς κανείς δεν εξετάσει πώς τελικά εξελίχθηκε η ανάπτυξη, Αυτό είναι προβληματικό και δυστυχώς πολύ συνηθισμένο στον τομέα των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου. Ας ξεκινήσω λοιπόν με ένα απλό μήνυμα. Με κίνδυνο να είμαι παράτολμος ε, στις γενικεύσεις μου, ε, Εάν διαβάσετε τη μελέτη θα διαπιστώσετε ότι είναι ιδιαίτερα αναλυτική. Δεν ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω από μεγάλο όγκο στατιστικών ε, που να φαίνεται να αντιφάσκουν κιόλα. Θα ξεκινήσω λοιπόν με ένα απλό μήνυμα το οποίο είναι ότι εξ ορισμού εάν ε, εξαλείψετε τους δασμούς σε ουσιαστικά όλες τις εισαγωγές, θα αφαιρέσετε και όλα, τα δασμολογικά έσοδα από τις εισαγωγές ε, από τις χώρες εταίρους σας. Και το εμπόριο που θα μεταφερθεί από τομείς σε μη απελευθερωμένους σε απελευθερωμένους τομείς σημαίνει ότι στο τέλος μπορεί να αυξηθούν τα έσοδα κατά την περίοδο εφαρμογής, διότι όσο χαμηλώνουν οι δασμοί, αυξάνονται οι εισαγωγές και έτσι αυξάνεται, αυξάνονται τα συνολικά έσοδα. Τελικά όμως οι δασμοί θα μηδενιστούν και έτσι, τα αντίστοιχα έσοδα επίσης θα είναι μηδενικά. Και γι' αυτό η απελευθέρωση του εμπορίου διαφέρει από άλλες μορφές απελευθέρωσης είτε στο πλαίσιο προγραμμάτων ε, διαφρωτικής ε, προσαρμογής, είτε στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων όπου η απελευθέρωση μπορεί να μην οδηγήσει σε μηδενισμό και έτσι να μην υπάρξει αλλαγή του εμπορίου, διότι η απελευθέρωση θα ισχύει για όλους τους εμπορικούς εταίρους. Το άλλο σημαντικό μήνυμα είναι ότι αυτή η απώλεια εσόδων μπορεί να είναι πολύ σοβαρή για κάποιες χώρες. Νομίζω ότι σε διάφορες μελέτες έχουν ε, εκφραστεί πολλές υπερβολές σχετικά με τις απώλειες κάποιων χωρών ΑΚΕ. Αντίστροφα όμως έχει υπάρξει εφησυχασμός ε, σχετικά με τον τρόπο που μπορούν να αποκτηθούν ε, εναλλακτικές ε, πηγές εσόδων. Μία από τις λίγες μελέτες που εξέτασαν τι έγινε στην πραγματικότητα όταν κράτη απελευθέρωσαν το εμπόριο, εξέτασε η μελέτη αυτή 115 χώρες κατά τη διάρκεια 100 ετών και τα αποτελέσματα είναι συγκλονιστικά. Οι πλούσιες ε, χώρες και χώρες μεσαίου εισοδήματος ε, σε μεγάλο βαθμό ήταν επιτυχής ε, κατά την αντικατάσταση των εσόδων, διότι αυξήσαν άλλες πηγές φορολόγησης, αλλά οι φτωχές χώρες δεν τα κατάφεραν εξίσου καλά για κάθε δολάριο που χάθηκε, μόνο 37 cents ε, έχουν ανακτηθεί από εναλλακτικέ ε, πηγέ φορολόγηση. Ακόμα και ελάχιστες μειώσεις ε, σόδων κρατικών ως αποτέλεσμα συμφωνιών μπορούν να αποτελέσουν σημαντικές προκλήσεις για τη χρηματοδότηση των χωρών αυτών. Και νομίζω ότι το τμήμα αυτό της μελέτης σχετίζεται πολύ με τη συζήτηση που μόλις είχαμε σχετικά με τα επίπεδα βοήθειας. Να προχωρήσω σε πιο αναλυτικά συμπεράσματα. Είναι γεγονός ότι οι επιπτώσεις στα έσοδα ε, είναι πολύ συγκεκριμένες όσον αφορά κάθε χώρα και κάθε ε, συμφωνία. Υπάρχει πολύ ευρύ φάσμα ε, στον βαθμό από τον οποίο εξαρτώνται από τα έσοδα που προέρχονται από δασμούς ε, εισαγωγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ευρύ φάσμα όσον αφορά το βαθμό που εξαρτώνται από τους δασμούς ως πηγή κρατικών εσόδων. Η υποσαχάρια Αφρική συνολικά εξαρτάται περισσότερο από τα έσοδα αυτά από ότι άλλες αναπτυσσόμενες περιφέρειες, αλλά ακόμα εντό ε, της υποσαχάριας Αφρικής υπάρχουν τεράστιες διαφορές ανάμεσα στις διάφορες χώρες. Και γενικά υπάρχει μεγάλη διαφορά και σε άλλες περιοχές της Και φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πάντα η πιο σημαντική πηγή εισαγωγών. Ε, ακόμα και στην Καραϊδική και τον Ειρηνικό υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση ε, ο Ειρηνικός ε, εισάγει πολύ από τη Ιαπωνία, η Καραϊβική από την Αμερική. Αλλά ε, η εξάρτηση από, τις, από τους δασμούς είναι μεγαλύτερη από ό,τι στην Αφρική, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και πάλι υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές. Άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι όλες από τις 17 μελέτε που εξετάσαμε, που συμπεριλαμβάνουν και τι μελέτε αντικτύπου για τη βιωσιμότητα που έχουν δημοσιευτεί, οι προβλέψεις που έγιναν Προτού να είναι γνωστά τα τελικά αποτελέσματα των συμφωνιών εταιρική σχέση και προτού να είναι γνωστό σε για ποια προϊόντα θα υπάρξει απελευθέρωση και πότε, δεν δείχνουν και την ταχύτητα με την οποία θα ε, απολεσθούν τα έσοδα αυτά, ούτε τα συνολικά ποσά. Η ε, διάρκεια εφαρμογής των συμφωνιών εταιρικής σχέσης ποικίλει από 8 σε 25 χρόνια σε κάποιες περιπτώσεις. Καμία χώρα ΑΚΕ δεν δημοσιεύει στοιχεία σχετικά με το πόσα έσοδα έχει από εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάτι που επαναλαμβάνεται συχνά είναι ότι δεν μπορεί να χάσει κανείς περισσότερα έσοδα από ό,τι έχει κάποια συγκεκριμένη στιγμή. Λαμβάνοντας υπόψη όμως τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή των συμφωνιών, πιστεύουμε ότι το μεγαλύτερο πλήγμα όσον αφορά την απώλεια εσόδων ε, θα φανεί ε, περίπου στο μέσο της διάρκειας εφαρμογής ε, της κάθε συμφωνίας εταιρικής σχέσης, δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις μετά από τέσσερα χρόνια ήδη. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι τέσσερα ή οχτώ χρόνια είναι πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σαν το ε, ανοιγοκλείσιμο του ματιού. Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις ε, στο τελωνιακό σύστημα. δεν μπορώ να τονίσω αρκετά το πόσο μακρύς και δύσκολος είναι ο δρόμος ε, ε, ε, μεταβολής προς μια βιώσιμη φορολογική βάση σε εποχές απελευθέρωσης. Ούτε μπορώ να τονίσω αρκετά το πόση λίγη βοήθεια παρέχεται για τις μεταρρυθμίσεις των δημοσιονομικών και τελωνιακών συστημάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλος χορηγός της βοήθειας για το εμπόριο. Το 1 τρίτο περίπου όλης της βοήθειας που δόθηκε ε, προερχόταν από ε, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τα κράτη-μέλη. Σχετικά μικρό ποσοστό όμως ε, έχει ταξινομηθεί στις κατηγορίες του ΟΣΑ που σχετίζονται περισσότερο με την ε, μεταρρύθμιση φορολογικών συστημάτων. Το σύστημα του ΟΣΑ βέβαια δεν είναι τέλειο, απέχει πολύ από τον ανετέλειο. Οι χορηγοί κατηγοριοποιούν τη βοήθειά τους ανάλογα με τον τίτλο που θεωρούν πιο κατάλληλο και φυσικά μπορεί κάποια προγράμματα να καλύπτουν διάφορες κατηγορίες και που να κατηγοριοποιούνται σε άλλη κατηγορία ε, από αυτή που σχετίζεται περισσότερο με τις θελονικές μεταρρυθμίσεις, ε, που είναι οι προσαρμογές που σχετίζονται με το εμπόριο. Αλλά, ακόμα και με αυτή την επιφύλαξη, φαίνονται ε, ελάχιστα τα ποσά που δίδονται στον τομέα αυτών και πρέπει να πω ότι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σχεδόν ο μόνος χορηγό ε, βοήθειας στον τομέα αυτών. Ε, στη μελέτη θα διαπιστώσετε ότι έχουμε εντοπίσει για όλες τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία την κατηγορία, τις κατηγορίες μάλλον, που σχετίζονται με τις μεταρρυθμίσεις ε, στον φορολογικό τομέα. Και θα επισημάνω ένα στοιχείο εδώ. Εξετάσαμε περίοδο 9 ετίας και εξετάσαμε όχι αποκλειστικά όμως, κυρίως όμως 16 χώρες που φαίνονται απριόρι να βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο ή πολύ υψηλό κίνδυνο όσον αφορά την απώλεια σημαντικού τμήματος των κρατικών εσόδων ε, λόγω της εφαρμογής συμφωνίας εταιρικής σχέσης. Από τις 16 αυτές χώρες και σε διάρκεια 9 ετών, μόνο τρεις είχαν λάβει βοήθεια προσαρμογής που σχετίζεται με το εμπόριο ε, ύψους πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια. Στην άλλη άκρη της κλίμακας, σε τρεις χώρες δεν είχαν λάβει τίποτα, ενώ άλλες τρεις είχαν λάβει λιγότερο από 10.000 ευρώ το χρόνο. Ε, που είναι ε, γελίο ποσό. Οι υπόλοιπε είχαν λάβει κατά μέσο όρο λιγότερο από 200.000 δολάρια το χρόνο. Θα ήθελα τώρα να τονίσω ότι οι στατιστικές αυτές είναι οι βέλτιστες διαθέσιμες αυτή τη στιγμή. Δεν είμαστε σε θέση ε, να Έχουμε αντίλογο όσον αφορά τον τρόπο που οι χορηγοί κατηγοριοποιούν τη βοήθειά τους. Επίσης, ε, ε, συχνά δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Ε, κάποια προγράμματα βοήθειας μπορεί να έχουν μπει σε διαφορετική κατηγορία. Θα ήταν όμως υπερβαλλικά αισιόδοξο δεδομένων των περιορισμένων ροών στην κατηγορία που σχετίζεται περισσότερο με τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις, ε, να θεωρήσουμε ότι οι πόροι που διατίθενται αυτή τη στιγμή ε, αρκούν για τις, αρκούν για τις ανάγκες. Και μάλιστα μπορεί ήδη σε τέσσερα χρόνια να έχουμε την ε, στιγμή των μεγαλύτερων απολειών για κάποιες χώρες. Με βάση λοιπόν αυτές τις αναλύσεις ε, που ε, παρουσιάζονται πολύ πιο αναλυτικά στο έγγραφο, έχουμε υποβάλει έξι συστάσεις, τις οποίες θα συνοψίσω εδώ. Με βάση έναν τίτλο και τις έχω χωρίσει μάλιστα σε τρία βήματα. Ε, ο βασικός τίτλος λοιπόν ε, που Το βασικό θέμα είναι ότι η κοινοβουλευτική συνέλευση βρίσκεται σε πολύ καλή θέση ώστε να ασκήσει πίεση για να χρησιμοποιηθεί η βοήθεια που δίνεται στο πλαίσιο Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΚΕ σε χώρες ε, που προσπαθούν να εφαρμόσουν ε, δημοσιονομικές και τελωνικές μεταρρυθμίσεις. Θα πρέπει να ληφθεί τέτοια απόφαση. Τέτοιες μεταρρυθμίσεις ε, συνεπάγονται τροποποιήσεις, μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται πολύ κοντά στον πυρήνα των πολιτικών που θεωρούνται αρμοδιότητα των κυρίαρχων κρατών. Δεν έχουν διάθεση όλες οι χώρες να μεταρρυθμίσουν τους τομείς αυτούς. ενώ παράλληλα καμία εξωτερική βοήθεια δεν θα οδηγήσει σε ε, ικανοποιητικά αποτελέσματα αν το θέμα αυτό δεν αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα. Η μεταρρύθμιση του φορολογικού είναι μακροπρόθεσμη διαδικασία, χρειάζεται τουλάχιστον μία δεκαετία και ε, απαιτούνται βήματα προς πολλές κατευθύνσεις και από τους χορηγούς και από τους δικαιούχους. Όπως συζητήθηκε και πριν, λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει κοινή οικειοποίηση ενός τέτοιου προγράμμα, προγράμματος ε, εάν θέλουμε να υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα επιτυχίας. Θα πρέπει λοιπόν ε, να ε, διαπιστωθεί καταρχάς ε, που θα είναι οι μεγαλύτερες απώλειες στην αρχή. Οι περισσότερες προβλέψεις, όπως σας είπα, έγιναν προτού να συναυθούν οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης, προτού να υπάρξει συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα και προτού να υπάρχουν στοιχεία σχετικά με το ύψος των εσόδων που συλλέγονται αυτή τη στιγμή ε, πάνω στις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι όπως σας είπα δεν μπορεί να χάσει κανείς ε, περισσότερα έσοδα από αυτά που ήδη συγκεντρώνει. Και ε, τα πραγματικά έσοδα είναι πάντα πιο χαμηλά από αυτά που έχουν υπολογιστεί, διότι υπάρχουν εξαιρέσεις, υπάρχουν αφορολόγητα προϊόντα κλπ. Οι μελέτες λοιπόν αποτελούν ε, κάποια καθοδήγηση σχετικά με το από πού θα πρέπει να ξεκινήσει κανείς. Ε, ξέρουμε έτσι για ποιες χώρες υπάρχουν κάποια εκ των προτέρων ε, στοιχεία που δείχνουν ότι κινδυνεύουν περισσότερο επειδή σημαντικό τμήμα των κρατικών τους εσόδων προέρχεται από τους δασμούς εισαγωγών και επειδή η διάρκεια εφαρμογής είναι σχετικά σύντομη της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης. Αφού λοιπόν ε, ε, διαπιστωθεί ποιες χώρες ε, βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλες οι συμφωνίες εταιρική σχέσης, ώστε να παρασχεθεί μεταβατική βοήθεια όπου αυτή είναι απαραίτητη και πιο μακροπρόθεσμα να υποστηριχθούν οι μεταρρυθμίσεις στο δημοσιονομικό και φορολογικό τομέα στις χώρες ΑΚΕ που έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν τέτοιες μεταρρυθμίσεις. Γενικά οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης ε, έχουν αρκετά γενική διατύπωση όσον αφορά τις ε, σχετικές συστάσεις. Οι πιο πρόσφατες ε, συμφωνίες είναι πιο συγκεκριμένες και στο παράρτημα έχουμε συμπεριλάβει τα σχετικά τμήματα από κάθε συμφωνία εταιρικής σχέσης. Κάποιες συμφωνίες εταιρικής σχέσης αναφέρουν ε, συγκεκριμένα την ε, στήριξη που δίνεται για ε, μεταρρυθμίσεις στον δημοσιονομικό και φορολογικό τομέα. Καμία τέτοια συμφωνία δεν αποκλεί να δοθεί βοήθεια για τέτοιες μεταρρυθμίσεις. Το θέμα με τις γενικές διατυπώσει είναι ότι είναι γενικές, ότι μπορούν να καλύψουν οτιδήποτε. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία συμφωνία εταιρική σχέσης που να μην επιτρέπει νομική βάση για τις χώρες που το επιθυμούν, ώστε τμήμα της ε, βοήθεια που χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δοθεί στην μακροπρόθεσμη διαδικασία για τροποποίηση της φορολογικής βάσης που θα είναι απαραίτητο να γίνει λόγω της ε, συμφωνία εταιρική σχέσης ε, και που θα είναι και απαραίτητη διότι φαίνεται ότι ε, μετακινούμαστε σε μια περιοχή εμπορικής απελευθέρωσης. Και τέλος έχουμε τη διαδικασία εκ των υστέρων παρακολούθησης. Ο λόγος που δεν μπορώ να σας πω τι επιτυχίες υπήρξαν στο παρελθόν κατά την υποκατάσταση της φορολογικής βάσης είναι ότι έχουμε σημαντικό κενό στις γνώσεις μας. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι επιτυχία θα έχουν οι συμβαλόμενοι των συμφωνιών αυτών ε, στην υποκατάσταση των φορολογικών εσόδων, διότι τώρα μόλις ξεκινάμε, αλλά είχαμε συμφωνίες ελεύθερο εμπορίου επί πολλά χρόνια και κατά την εξέταση 144 μελετών των ε, συμφωνιών ε, ελεύθερου εμπορίου κατά τα τελευταία 50 χρόνια, στη μελέτη αυτή δεν διαπιστώθηκε ούτε μία περίπτωση σωστής ανάλυσης σχετικά με το τι είχε γίνει. Στην περίπτωση της ΑΚΕ, η παρακολούθηση, η εκ παρακολούθηση θα πρέπει να εξετάσει τις επιπτώσεις της ανακατανομής στα κρατικά έσοδα συνολικά. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο φαίνεται να ε, πιστεύει ότι οι χώρες οι πιο επιτυχείς τα κατάφεραν ε, με φόρους κατανάλωσης, ε, είτε ε, ΦΠΑ είτε φόρο επί των πολίσεων. Είναι κάπως απίθανο αυτή η φόροι να ε, έχουν ακριβώς το ίδιο ύψος ε, με τους δασμούς. Δηλαδή, μπορεί οι φόροι σε κάποια προϊόντα να αυξηθούν, σε άλλα να μειωθούν. Άλλωστε, οι διαφορετικές χώρες ε, έχουν και διαφορετικό καλάθι κατανάλωσης. Είναι πολύ σημαντικό να διαπιστώσουμε εάν οι τιμές των αγαθών που απευθύνονται σε πιο ευάλωτες ομάδες αυξάνονται ή μειώνονται. Στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πρέπει η παρακολούθηση να γίνει για να διασφαλιστεί το ότι γίνονται σωστά βήματα με κοινή δέσμευση της ΑΚΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα ε, εγγενές στην όλη διαδικασία ΑΚΕ. Και έτσι επανέρχομαι στην αρχική μου θέση ότι εάν εξαλειφθούν οι δασμοί στις εισαγωγές, χάνει κανείς τα έσοδα από τις εισαγωγές ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς ε, και ε, εμπορικών συναλλαγών από κάποιες άλλες πηγές. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να αποτελέσει σημαντική ανησυχία όσον αφορά τις εμπορικές ροές που παρακολουθεί η κοινή κοινοβουλευτική συνέλευση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you, Ευχαριστούμε κύριε Στίβενς για την τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Τώρα το λόγο έχουν τα μέλη της Επιτροπής μας εδώ που θέλουν να κάνουν σχόλια ή να υποβάλουν ερωτήσεις. Παρακαλώ. Η Νότια Αφρική. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση. του καθηγητού Στίβενς, έτσι. Θέλω να προτείνω πάλι ότι για να προχωρήσουμε στο μέλλον όσον αφορά την παγίωση ισότιμων σχέσεων και εταιρικών σχέσεων των χωρών και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να μην αποκλείουμε κανέναν. Ίσως αυτό που λέτε ότι οι πληροφορίες δεν υπάρχουν ή δεν είναι γνωστές, κάποιοι καθηγητές από τον Ιρωνικό ή από την Αφρική να έχουν διαφορετική άποψη από σας. Τώρα διορθώστε με αν κάνω λάθος. Χρειάζεται μια πιο βαθιά επιστημονική ανάλυση όσον αφορά τον αντίκτυπο της ελευθέρωσης του εμπορίου τις τελευταίες τρεις με τέσσερις δεκαετίες. Οι συστάσεις σας πρέπει να περάσουν από αυτό αυτά ακριβώς τα γυαλιά της ανάλυσης αυτής που σας λέω. Αλλιώς θα υπάρξουν χαμένοι. Και μιλάω για αυτή την επιστημονική ανάλυση, γιατί ιστορικά αυτούς τους χαμένους θα τους βρείτε στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, στις χώρες εκείνες που δεν έχουν οικονομική ισχύ. Οι χαμένοι θα είναι αυτές οι φτωχές μάζες μέσα στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Οι χαμένοι θα είναι αυτοί οι φτωχοί εργαζόμενοι ε, τους οποίους εκμεταλλεύονται άλλοι μέσω της ελευθέρωσης που δημιουργεί ανεργία. Και υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Στη Γεωργία, για παράδειγμα, πολλά. Τώρα, θα συμφωνήσω μεν μαζί σας, αλλά δεν νομίζω ότι τονίσατε παρκώς ότι χαμένοι είναι οι φτωχές χώρες. οι πιο φτωχοί στις υποανάπτυκτες ή στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες καταστρέφονται οι θέσεις απασχόλησης. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι το εξή. Αναφερθήκατε σε χώρες που είναι απόλυτα εξαρτημένες από τους δασμούς. Τους χρειάζονται γιατί αυτό είναι το εισόδημά τους, τα εσοδά τους. Συμφωνώ μαζί σας. Αλλά σε χρόνο σημαντικό είναι να δούμε ότι όταν μιλάμε για μεταβατικά μέτρα υπό τη μορφή βοήθειας, για να αντισταθμίσει το, τα έσοδα που θα χαθούν, να ξέρουμε ότι οι απώλειες θα είναι μακροχρόνιες και σημαντικές. Οι περισσότερες φτωχές χώρες χρησιμοποιούν σαν κοινωνικό εισόδημα τους δασμούς. Σε αυτό συμφωνώ μαζί σας. Τρίτον, στήριξη στις μεταρρυθμίσεις στις χώρες ΑΚΕ. Δεν ξέρω εσείς πώς και σε ποιο πλαίσιο βλέπετε τις χώρες αυτές και Τις χώρες αυτές οι οποίες έχουν δεσμευτεί για μεταρρυθμίσεις και στα τελωνία. Κύριε καθηγητά Στίβενς, επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στις χώρες μας, σήμερα έχουμε ε, υπηρεσίες ε, πιστοτικές. Είναι υπηρεσίες αξιολόγησης, οι οποίες υποβαθμίζουν τη χώρα σας και χρησιμοποιούν τις μεταρρυθμίσεις σαν καθοριστικό παράγοντα για να μας πούνε αν θα μας υποβαθμίσουν ή θα μας αναβαθμίσουν ως χώρα. Λένε πρώτο πρέπει να γίνει μεταρρύθμιση, δεύτερον πρέπει να μειώσετε τις δαπάνες, τέλος πάντων να βάλετε κάποια ισορροπία στις δαπάνες. Ιστορικά όμως μιλώντας, ότι όλα αυτά αποδυναμώνουν τους φτωχούς τελικά. Γιατί όταν το κράτος θα μειώσει τις δαπάνες, θα μειώσει τις δαπάνες στις κοινωνικές υπηρεσίες, στην υγεία, στην εκπαίδευση κλπ. Όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε και θα συζητήσουμε είναι αλληλένδετα μεταξύ τους και όταν τα συζητάμε πρέπει να τα συζητάμε συνολικά γιατί ακριβώς είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Θα σταματήσω εδώ, γιατί σας είπα τα πιο βασικά που ήθελα να πω. Αλλά και πάλι, πώς θα μετρήσουμε την δέσμευση κάποια για μεταβατικά μέτρα που θα εφαρμόσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ουινέα. Σας ευχαριστώ, πράδρα το θέμα που είναι η αντιμετώπιση των προκλήσεων στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες βάσει του ελεύθερου εμπορίου. Αυτό είναι το θέμα μας. Η εξαίρετη παρουσίαση που ακούσαμε τοποθετείται στην υπόθεση όπου οι χώρες έχουν την ικανότητα να αλλάξουν. οι χώρες που έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν, συμφωνώ μαζί σας καθηγητά Στίβενς, πρέπει να προχωρήσουν σε φορολογικές και τολωνιακές μεταρρυθμίσεις, πολύ σημαντικές για να εξασφαλίσουν εισόδημα. Αλλά κύριε καθηγητά, μια χώρα που δεν έχει τέτοια δυνατότητα, πώς θα κάνει, τι θα κάνει. Η πρώτη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας, η δυσκολία, είναι ακριβώς να έχουν αυτή τη δυνατότητα, αυτή την ευκαιρία να κάνουν τις αλλαγές. Όταν ανοίξετε την αγορά σας, δεν έχετε δυνατότητα, την ανοίγετε την αγορά σας για την παραγωγή αυτού που έχετε δυνατότητα. Τι θα γίνει όμως με τις ε, επιτόπου δυνατότητες. Αυτές ασφιξιούν σαν αποτέλεσμα. Οπότε να λύσουμε τις δυσκολίες των ε, υποανάπτυξη χώρων σημαίνει να ενισχύσουμε πρώτα απ' όλα τη δικιά τους ικανότητα να παράγουν και να εμπορεύονται. Χρειάζεται λοιπόν να ενισχύσουμε την ικανότητά τους να εμπορεύονται, να συναλλάσσονται. Πολύ καλή η παρουσία, αλλά για χώρες που ήδη έχουν εμπορικές συναλλαγές και για να μην χάσουν έσοδα πρέπει να προχωρήσουν σε δημοσιονομικές και τελωνιακές μεταρρυθμίσεις. Σύμφωνοι. Θέλω φυσικά να ακούσω την αντίδραση του καθηγητή για αυτήν την πρόκληση στην οποία αναφέρθηκα, που είναι η ενίσχυση της ικανότητας παραγωγής των υπανάπτυξη χωρών. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρένα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Στίβενς για την παρουσίασή του. Πριν από λίγο είχα διαβάσει μια ανάλυση του South Center που ανέφερε ακριβώς τις ίδιες πραγματικότητες που αναφέρατε κι εσείς. Πρόκειται για εμπειρογνώμονες, για επιστήμονες από χώρες αφρικανικές που εκπώνησαν τις μελέτες αυτές και καταλήγουν στην ίδια διαπίστωση όσον αφορά την απώλεια εσόδων για τις συμφωνίες αυτές εταιρική σχέσης και μιλούν για τις απώλειες αυτές λέγοντας ότι αυτοί που χάνουν περισσότερο είναι ακριβώς οι πιο φτωχές χώρες. Γιατί όταν μπαίνουμε σε μια λογική συναλλαγών η μείωση των τελών δεν είναι για να εισάγουμε περισσότερο, είναι για να εξάγουμε περισσότερο. Οπότε το πρόβλημα, όπως πολύ σωστά λέτε, είναι ότι αν δεν έχετε την εξάγετε, αν δεν έχετε παραγωγή, αν δεν μπορείτε να πάτε εσείς προς την αγορά του άλλου, τότε μόνο απώλεια εισπράτεται από την μείωση των δασμών, γιατί μπαίνουν λιγότερα στη χώρα σας. Και πληρώνετε πιο ακριβά ότι μπαίνει. Οπότε πώς να προχωρήσετε. Αυτό που συζητήσαμε μέχρι τώρα είναι πώς να βοηθήσουμε να υπάρχουν μεταπημένα προϊόντα τα οποία ακριβώ μπορούν να εξαχθούν από τις χώρες σας. Συνεπώς ο καθηγητής φυσικά δεν μπορεί να λύσει όλα τα ζητήματα και να αναφερθεί σε όλα, αλλά αυτό που συζητάμε εδώ τώρα είναι ότι αν δεν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε εξαγωγή μεταπημένων προϊόντων, να μπούμε σε μία, το, να το να μπούμε τότε σε μία συμφωνία εταιρική σχέση μπορεί να αποτελεί μειονέκτημα. Για τις χώρες ΑΚΕ έχουμε και περιφερειακές συμφωνίες, τουλάχιστον η Ευρώπη αυτό προσπαθεί να πετύχει, όπου έχουμε μία ή δύο χώρες μεσαίων εσόδων, ενώ οι υπόλοιπε χώρες είναι λιγότερο πλούσιες και που πραγματικά θα τα χάνανε όλα. Έχουν ήδη προτιμησιακή πρόσβαση στην Ευρώπη, οπότε δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα από δασμούς, αλλά θα χάσουν όσον αφορά ε, τα έσοδά τους και τις αγωγές τους. Οπότε βάσει της μελέτης σας κύριε καθηγητά θέλω να ρωτήσω πιστεύετε ότι πρέπει να συμβουλέψουμε τις χώρες εταίρους να μπουν στη λογική των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών έτσι όπως προτείνονται σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η προσωπική μου γνώμη είναι πως όχι. Σας το εξήγησα ήδη. Αλλά αν ένας επιστήμονας πει το ίδιο, ίσως αυτό να βαρύνει πολύ περισσότερο από ό,τι όταν το λέει ένας πολιτικός. Okay, so thanks for these interesting questions. If... Εάν δεν έχει ερωτήσεις, ναι, παρακαλώ. Εγώ. Ευχαριστώ κυρία Συμπρόεδρε. Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστούμε για τη σαφήνεια της εργασίας σας. Κύριε Καθηγητά, αν σας παρακολουθήσαμε σωστά, βασιστήκατε σε πάνω από 60 μελέτες. Και αυτό που θα θέλαμε να γνωρίζουμε είναι για τις χώρες που όντως ε, προχώρησαν στην κατάργηση των δασμολογικών ε, φραγμών, ποιες είναι οι περιφέρειες ή οι χώρες που κατάφεραν να σταθεροποιήσουν τα έσοδά τους. Πιστεύω ότι ε, Πολύ θα θέλαμε να έχουμε περισσότερε λεπτομέρειε. Υπάρχουν κάποια πρότυπα, κάποιε περιφέρειε ή κάποιε χώρε που τα κατάφεραν αφού προχώρησαν στην κατάργηση των δασμολογικών φραγμών να σταθεροποιήσουν τα, τα έσοδά του. Ευχαριστώ. I'm really sorry, but I have to leave and... Λυπούμε, αλλά πρέπει να φύγω, οπότε θα ε, δώσω τώρα την Προεδρία στη Συμπρόεδρο. Thank you. Thank you very much, uh, Laura Ferrara. Uh, Ευχαριστώ. Is there anybody else or shall I give it the... Ευχαριστώ. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο να κάνει άλλος ερώτηση. Ή να δώσω το λόγο στον εισηγητή για να απαντήσει στις ερωτήσεις που θέσατε. Και εγώ ως πρόεδρος ε, διαρωτώ αν μπορώ και εγώ να θέσω μια ερώτηση. Είδα τις στατιστικές, εγώ είμαι από την Κένια και διαπίστωσα ότι οι περισσότερες μελέτες ε, χρονολογούνται από το 2006-2007. Διερωτώ με αν είναι ακόμα έγκυρα αυτά τα στοιχεία το 2017, γιατί έχουν γίνει πολλές αλλαγές σε όλες τις χώρες και η βάση εισόδων επί της οποίας έχουν γίνει αυτές οι μελέτες έχει αλλάξει. Διερωτώμε λοιπόν πόσο έγκυρα είναι αυτά τα στοιχεία σήμερα, μετά από τόσα χρόνια. You, have the floor, Mr. Μάλιστα κύριε Στίβεν, έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τα σχόλια σας, ε, τα δικά σας. Είναι αλήθεια ότι οι περισσότερες αυτές μελέτες είναι ήδη αρκετά ε, ξεπερασμένες και επίσης η, τα έσοδα των χωρών ε, είναι πολλά και διάφορα και διαφέρουν μεταξύ τους όπως βλέπετε από τα στοιχεία που μας στάνουν και το 2012 στο δεύτερο πίνακα. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτή τη στιγμή οδηγούμε στην ομίχλη χωρίς φωτοομίχλη. και μάλιστα τρέχουμε κιόλα. Και θα ήταν πολύ λογικό να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις μελέτες απλά για να εντοπίσουμε πώς θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε τα στοιχεία που έχουμε από το παρελθόν. Τώρα, αρκετοί ομιλητές αναφέρθηκαν στην ε, ανταπόκριση στις συμφωνίες ε, τις εμπορικές ανάμεσα στις πιο αναπτυγμένες και τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες εντός της ομάδας των χωρών ΑΚΕ. Για να μπορέσουμε να εστιάσουμε την προσοχή και να δώσουμε μια λεπτομερή ανάλυση μιας πτυχής ενός θέματος θα πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό και να μην κοιτάμε όλα τα στοιχεία. Αυτή η μελέτη δεν είναι μία γενική εικόνα των υπέρ και των κατά των εμπορικών συμφωνιών. Εστιάζεται και συγκεκριμένα στο πώς θα έπρεπε να προσαρμοστούμε στις επιπτώσεις στα έσοδα για τις χώρες που αποφάσισαν να μπουν σε τέτοιες ε, συμφωνίες. Εάν με ρωτούσατε αν ε, κατά τη γνώμη μια χώρα θα έπρεπε να το κάνει αυτό, εγώ έχω κάνει έρευνα σχετικά με αυτό το θέμα εδώ και 20 χρόνια και απλά να πατήσω στο Google τι έγραψα, για να, πατήστε μάλλον το Google για να δείτε τι έχω γράψει, για να καταλάβετε ποια είναι η γνώμη μου. Αυτό όμως η αυτή έκθεση δεν αφορά αυτό, αφορά το θέμα των εσόδων. Και κατανοώ τα όσα είπε ο εκπρόσωπος της Νότιας Αφρικής, ότι δηλαδή χρειάζεται να έχουμε μελετητές από όλη την ομάδα των Χρονακέ. εδώ πρόκειται για μια εξέταση των σχετικών μελετών όπου περιλαμβάνονται και συντάκτες ε, από τις χώρες ΑΚΕ. Όσον αφορά όμως τη συνέχεια των μελετών που πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνει, να υπάρξει, εκεί θα πρέπει όντως να συμμετέχουν τοπικοί ερευνητές. Τώρα, για το πώς προσαρμόστηκαν οι χώρες στην απώλεια των δασμολογικών τους εσόδων, θα σας πω κάτι που είναι κάπως ε, ε αλλά έχουμε το, το έκτο γράφημα στη σελίδα νομίζω 16, όπου μπορείτε να δείτε κάποια παραδείγματα των επιπτώσεων που έχουν εντοπιστεί σε ορισμένες χώρες. We've come across, there are cases in which quite poor countries have apparently seen tariff, seen government revenue in. Βλέπουμε, είδαν λοιπόν τελικά ότι τα έσοδα των, τα κρατικά αυξήθηκαν στη διάρκεια της απελευθέρωσης και της μετα, φορολογικής μεταρρύθμισης. Το μόνο ίσως πρόβλημα που υπήρξε υποψιάζομαι, αλλά δεν είμαι βέβαιος, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η απελευθέρωση έγινε στο πλαίσιο είτε του πολυμερούς γύρου είτε των διευθυντικών προσαρμογών. Οπότε δεν ήταν απαραίτητο ε, ε, εκμυδένιση των φορολογικών δασμών. Και βεβαίω, εάν μειώσει τις δασμού από το 25% ας πούμε στο 8%, τότε μάλλον θα δεις αύξηση στα έσοδα λόγω του όγκου των εισαγωγών που θα αυξηθεί και άρα θα έχεις ναι μεν λιγότερο φόρο ανά ε, εισαγωγή αλλά έχεις πάλι περισσότερα έσοδα γιατί εισάγονται περισσότερα λοιπόν το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να φτάσουν υποτίθεται οι δασμοί στο μηδέν μέχρι το τέλος της περίοδου εφαρμογής και γι' αυτό λίγες αποδείξεις που έχουμε για την επιτυχία ή μη των χωρών που προσαρμόστηκαν ε, μετά από τις ε, δασμολογικές μεταρρυθμίσεις δεν μπορούν πραγματικά να χρησιμεύσουν ως ε, γνώμονας για τους συνυπογράφονται σε συμφωνίες ε, εμπορίου. Τώρα, εγώ επίσης δεν ήθελα να εντοπίσω κριτήρια για να δούμε κατά πόσο μια χώρα είναι όντως ε, προσιλωμένη σε αυτό που έχει συμπογράψει όχι. Για οποιοδήποτε πολιτικό, το να αλλάξει κανείς τη φορολογία του είναι πολιτικός, πολύ επικίνδυνο πράγμα. Οπότε, δεν είναι διόλου σίγουρο ότι κάθε χώρα θέλει πραγματικά να αρχίσει μια τέτοια ιστορία ε, βάθρων ε, ε, μεταρρύθμισης Όμως, αν απόφαση ότι όντως θέλει να το κάνει, το επιχείρημα εδώ είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στηρίξει μια τέτοια προσπάθεια. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Και τώρα να δώσω το λόγο για μερικά λεπτά στον εκπρόσωπο της Επιτροπής και ίσως να μπορούσατε και εσείς να απαντήσετε στις ε, ερωτήσεις που ετέθησαν. Η μείωση των δασμών μειώνει τα κρατικά έσοδα για τις κυβερνήσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει χαμηλότερες τιμές και ε, για τις εταιρείες που εισάγουν ανταλλακτικά και χαμηλότερες τιμές άρα για τους καταναλωτές. Ε, η μείωση των ε, κρατικών εσόδων δεν θα αργοπορήσει ως συνέπεια των πολύ χαμηλότερων περιορισμών των δασμών από τις χώρες και από ό,τι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εμπορικέ συμφωνίες θα προωθήσουν την τοπική οικονομία ως συνέπεια Έχετε λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να απαντήσω μετά από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στα σχόλια που ακούστηκαν. Δεν θα αξιολογήσω την έκθεση, αλλά θέλω να πω και εγώ τι κάνουμε από πλευράς Κομισιών σε συνεργασία με τους εταίρους μας για να αντιμετωπίσουμε ορισμένε από τις προκλήσεις που αναφέρθηκαν. Καταρχάς, θέλω να υπογραμμίσω ότι συμφωνώ με το πόρισμα της μελέτης που λέει ότι Απαιτείται στήριξη της, ε, ε της δημοσιονομικής ε, ενίσχυσης της χρηματοοικονομικής στήριξης ε, για τους ε, εταίρους μας με τις συμφωνίες εικόνων εταιρικής Η βοήθεια για το εμπόριο ουσιαστικά βασίζεται στη ζήτηση, πρέπει να σας πω. Δηλαδή δεν θα επιβάλλει κομισιόν στις χώρες εταίρους βοήθεια που δεν τη ζητάνε. Και επομένως η βοήθεια για το εμπόριο βασίζεται σε αξιολόγηση των αναγκών στις χώρες επιτόπου. Αν υπάρχει ανάγκη κάποιων μέτρων εμπορικής προσαρμογής, αυτό μπορεί να φύγει στο γεγονός πολύ απλά ότι δεν υπήρξε ακόμα απελευθέρωση. Όταν μιλάμε λοιπόν για χώρες οικονομικής θερικής σχέσης, πρέπει στην Αφρική για παράδειγμα να δούμε ποιος είναι στις συμφωνίες και ποιος ετείται ε, εδώ και χρόνια. Λίγες είναι οι χώρες, ε, τέσσερις τον θυμώ. Η Ζιμπάμπουε ξεκίνησε πολύ πρόσφατα ε, την, κάποιες αλλαγές. Επομένως, αφού δεν υπάρχει δημοσιονομικό αντίκτυπος, είναι λογικό να μην υπάρχουν αντισταθμιστικά μέτρα. Σε ό,τι την αρχική και τελική παρατήρηση το μου καθηγητού. Λέτε ότι σωστικά θα χαθούν όλα τα εμπορικά έσοδα. Διαφωνώ μαζί σας σε όλες τις ΕΠΑ. Οι χώρες εταίροι κατάφεραν να προστατεύσουν μέχρι το 20% των δασμών και αυτό σημαίνει ότι έχουν προστατεύσει και τα, τις γραμμές αυτές που είναι ευαίσθητες. Δεν πάνε τα πράγματα όπως τα λέτε. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. αλκοόλ, αυτοκίνητα και τα λοιπά. Πρώτα ευαίσθητα δηλαδή δείχνουν ότι δεν επηρεάζονται τα κρατικά έσοδα τόσο πολύ. Σε ό,τι αφορά, αφού κλείσω την παρένθεση, την παρακολούθηση και το τι κάνουμε για να παρακολουθούμε το δημοσιονομικό αντίκτυπο και τι κάνουμε για να στηρίξουμε τις ε, δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις και απόλυση ε, εισοδήματος ε, ενδεχομένως. Σύμφωνα με τη συνήθεια μας πρακτική, διεξάγουμε μελέτες επιπτώσεων αφού δούμε, δούμε πώς πήγε η καθέπα για το Σάντεκα και τη Δυτική Αφρική, αυτό έχουμε κάνει ήδη. Βλέπετε τις σχετικές αναφορές στη μελέτη. Άρα δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες. Επίσης, κάνουμε περιοδικές αξιολογήσεις. Κάθε πέντε χρόνια ή κάτι τέτοιο. Ανάλογα με την ε, αίτηση. Έτσι μπορούμε να δούμε ποιες είναι οι προκλήσεις ε, στο τεφατή εισόδημα. Προβλέπουμε μια τέτοια μελέτη για την Ανατολική και Δυτική Αφρική το 2018 και για τον Ειρηνικό το 2019. Για την κάτι ακόμα. Οι κοινοί φορείς των ΕΠΑ που παρακολουθούν την εφαρμογή είναι εκεί για να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε πρόκληση προκύψει και σε ό,τι αφορά τι απώλειε εισοδήματο. Μέχρι στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάθε ΕΠΑ έχει αναλάβει τη δέσμευση να αντισταθμίσει την καθαρή εισοδηματική απώλεια. Δεν έχουμε λάβει μέχρι τώρα κανένα αίτημα αντιστάθμισης, αποζημίωσης. Και αυτό γιατί η απελευθέρωση Ε, γίνεται σταδιακά. We, we are ready to support this. Εμείς είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις, αλλά τις φορολογικές μάλλον μεταρρυθμίσεις, αυτό θα πρέπει να βασίζεται στη ζήτηση. Ό,τι αφορά τώρα τις έπατε που ισχύουν ε, από παλιά, 2008, με την Καραϊβική, με PNG, από το 2011, Ανατολική Αφρική, από το 2012, εδώ δεν έχουμε στιγμή ε, εντοπίσει σοβαρέ εισοδηματικέ απώλειε, γι' αυτό και δεν στήθηκε και κάποια υποστήριξη για την Καραϊβική. Ανακοίνωσε στην τελευταία συνάντηση, λίγου μήνε πριν ε, δηλαδή, ότι θα κάνουν μια μελέτη για το δημοσιονομικό αντίκτυπο τη συμφωνία ε, οικονομική και Εταιρική Σχέση και θα ξέρουμε περισσότερα στου επόμενου μήνε. Αυτέ είναι ευκαιρίε Να δούμε από κοινού με τους εταίρους μας τι προβλήματα υπάρχουν και πώς μπορούμε να τους υποστηρίξουμε, είτε με τη μορφή ε, μια διαδικασίας μεταρρύθμισης, είτε με τη μορφή αποζημίωση αντιστάθμισης της καθαρής οδηματικής απώλειας. Είναι σημαντικό να σημειώσω, το είπε και η κυρία Συμπρόεδρος, ότι η μείωση των, ε, η απώλεια των ε, εισαγωγικών δασμών αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει μείωση του συνολικού ΑΕΠ θα υπάρξει τόνος οικονομικών δραστηριοτήτων και όλες οι μελέτες που έχουμε διεξαγάγει για τον αντίκτυπο των ΕΠΑ δείχνει ότι θα συμβεί αυτό. Όπως πιο πρόσφατα με τη ΣΑΝΤΕΚ. Είδαμε εκεί ότι οι ισοδηματικές απώλειες θα είναι περιθωριακές, κατά μέσο όρο 0,51%. Συν το χρόνο πάντα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το συνολικό, συνολική, ο συνολικός αντίκτυπος θα είναι αρνητικός. Μάλιστα περιμένουμε αύξηση λόγω της οικονομικής ε, εταιρικής σχέσης. Και πολύ σωστά είπε και η συμπρόεδρος για τα εισαγόμενα ε, προϊόντα που επειδή είναι φθηνότερα συνεισφέρουν και αυτά σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγή, τοπική παραγωγή προϊόντων και μπορούν να αποφεληθούν από τις συναντρες τιμές βέβαια και καταναλωτές. Ξέρω ότι μακρηγόρησα, αλλά αν μου επιτρέπετε ένα ακόμη σημείο θέλω να αναφέρω, απαντώντας στην Μαρία Αρενά για τα μεταποιημένα προϊόντα. Θέλω να σας αναφέρω ένα παράδειγμα από τη Μαδαγασκάρη που είναι μία από τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές και εφαρμόζει ε, εδώ και κάποια χρόνια τώρα. Ακούσαμε ε, να γίνονται αναφορές και από τους ε, διάφορους κλάδους βιομηχανίες και από επιχείρησεις που λένε ότι αυτή η συμφωνία ουσιαστικά βοήθησε τους κλάδους να επιβιώσουν, που θα είχαν πτωχεύσει επιχειρήσεις κλωστοϊφαντουργικές για παράδειγμα και με ε, τις πρώτε ύλες ε, μπορούν να εξάγουν ε, αδασμολόγητα τις πρώτες ύλες στις αγορές της Ευρωπαϊκή Ένωση και μια συγκεκριμένη εταιρεία διατήρησε 2.000 απασχολούμενους ακριβώς για αυτό το λόγο. Παρότι ε, είπα, απέσυραν τα ωφέλη τους, τα πλεονεκτήματα μάλλον που έδιναν, μπορούμε να τα πούμε ίσως και σε μια άλλη περίσταση πιο διεξοδικά. Ευχαριστώ. Thank Any comment, last comment, Mr. Stevens? Ευχαριστούμε κύριε Στίβεν. Θέλετε να αντιδράσετε? Όχι? Ωραία. Τότε επιτρέψτε μου να συνεχίσω αγαπητοί συνάδελφοι. Κλείνει η συζήτηση για αυτό το θέμα. Um, as has become the custom now, we are... Ως ήθιστε, πάμε πάνω κάτω στην ημερήσια διάταξη, τι να κάνουμε. Η... ειδική για το θέμα της γαλάζιας οικονομίας, ευκαιρίες και προκλήσεις δεν είναι εδώ, γι' αυτό θα περάσουμε στο σημείο 8. Και θα επανέλθουμε στο 7 μετά, όταν θα έχουν έρθει οι εμπειρογνώμονες. Σημείο 8 λοιπόν. Είναι η συνέχεια που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ψήφισμα της κοινοβουλευτική Συνέλευσης και Ευρωπαϊκής για τις επιπτώσεις των ε, παράνομων ε, χρηματοπιστωτικών ροών στην ανάπτυξη. Το Δεκέμβριο του 2016 εγκρίναμε ένα ψήφισμα για τις επιπτώσεις αυτών ακριβώς των ροών ε, στις οικονομίες των χωρών ΑΚΕ. Με το ψήφισμα αυτό αναφέραμε την ανάγκη για διεθνείς προσπάθειες προκειμένου να καλυφθούν τα νομικά κενά, να υπάρξει περισσότερη διεθνή συνεργασία και διαφάνεια υπέρ της καταγραφής του φαινομένου αυτού. Πρέπει να γίνουν περισσότερα, να έχουμε εκθέσεις από κάθε χώρα χωριστά για τις δραστηριότητε των επιχειρήσεων και να καλυφθούν όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με παράνομα περιουσιακά στοιχεία. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας εξηγήσει τι συνέχεια δόθηκε στο ψήφισμα αυτό του σώματος. Παρακαλώ. Να χειροκροτήσουμε τον κύριο Στίβεν όμως, έτσι. Δεν το κάναμε πριν. Σας ευχαριστούμε. Ε, το παρέλειψα, λυπάμαι. Um, another hitch. Can we give you a five minutes break? Μπορούμε να διακόψουμε πέντε λεφτά. Ίσως για να πιούμε καφέ, το ξέχασα και αυτό. Και μετά θα επανέλθουμε στην αίθουσα. Γιατί δεν είναι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ο αρμόδιος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα μας μιλούσε για αυτό το θέμα. Ωραία. Οπότε, τεντωθείτε λιγάκι. Και να ξανάρθετε σε πέντε λεπτά, ελπίζοντας ότι θα έχουμε εδώ τον αρμόδιο.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 Right, right, members, just to get us back. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, να περάσουμε πάλι στην μεσιά διάταξη και στο θέμα που μας ε, απασχολεί και συγκεκριμένα ε, είναι το follow-up της Κομισιόν ε, στο ψήφισμα της Ένωσης Εκπροσώπησης Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΚΕ για τις παράνομες κανοικονομικές ροές σε ό,τι αφορά την ε, ανάπτυξη και βοήθεια. Το Δεκέμβριο του 2016 εγκρίναμε ένα ψήφισμα για τον αντίκτυπο των παράνομων χρηματοοικονομικών ε, ροών για την αναπτυξιακή χρηματοδότηση. Στο ψήφισμα αυτό, μεταξύ άλλων, τονίσαμε την ανάγκη για συντονισμένη διεθνή προσπάθεια ώστε να κλείσουν ε, τα νομικά κενά, να αναβαθμιστεί η διεθνή συνεργασία και να αυξηθεί δραστικά η διαφάνεια σε ό,τι αφορά την ε, ιδιοκτησία και τις χρηματοοικονομικές δωρές. Θα είναι περισσότερα για την ε, βελτίωση της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων αναχώρα, για τις ε, συγκεκριμένα τις πολυεθνικές εταιρείε και για την διευκόλυνση ανάκτηση των παράνομων εσόδων. Θα ήθελα να δώσω τώρα την Κομισιόν το λόγο να μας πει τι συνέχεια θα δώσει σε αυτό το ψήφισμα της συνέλευσής μας. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο, Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Χίμπερτ Πέρ και είμαι προϊστάμενος ε, του τομέα για την κινητοποίηση χώρων εισόδου στο πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξη αυτή η γενική διεύθυνση. Αν με επιτρέπετε, θα ήθελα να εστιάσω συγκεκριμένα στην εντολή της ΓΔ ΤΕΦΚΟ για τη συνέχεια, την παρακολούθηση και τις δράσεις που μπορούμε να αναλάβουμε για την αντιμετώπιση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών και τι μπορούμε να κάνουμε και στην, ε, στο πλαίσιο της εντολής μας για την αναπτυξιακή συνεργασία. Ότι δηλαδή ε, πρέπει να έχουμε παρέχουμε βοήθεια στις χώρες στη ΣΑΚΕ που έχουν πρόβλημα. Θα έρθει και ένας συνάδελφος από την Καμάθα Τάξουτ, ο οποίος θα σας μιλήσει πιο πολύ για τα ευρωπαϊκά φορολογικά ζητήματα. Έχω έναν συνάδελφο μαζί μου εδώ, από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΤΖΑΣΤ, τον κύριο Τόμας Λούγκβιστ. Θα σας ε, μιλήσει για ε, τους ε, τελικούς δικαιούς, πραγματικούς δικαιούχους ε, και το ξέπλυμα χρήματος και όλα αυτά στο πλαίσιο της αναπτυξιακής ατζέντας, του αναπτυξιακό θεματολογίου. Σε ό,τι αφορά τώρα τη διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη, συμφωνούμε απόλυτα με το περιεχόμενο του ψηφίσματος. Πολύ καλά αναφέρεται και επεξηγείται το μέγεθος των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών και τη σημασία που έχουν για την Ευρώπη, αλλά κυρίω για τι αναπτυσσόμενε χώρε και τι χώρε ΑΚΕ. Όπω γνωρίζουμε όλοι, αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο σε αναπτυσσόμενε χώρε. Και επειδή έχουμε την ε, δραστηριότητα αυτή της κινητοποίησης εγχώριων εισόδων στο πλαίσιο της διαδικασίας Αντίσα Μπέμπα. θέλουμε να πετύχουμε και να βελτιώσουμε την κινητοποίηση αυτή, αυτό θα πρέπει να το κάνουμε ε, αντιμετωπίζοντας και τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές. Πολύπλοκο το ζήτημα, με πολλές πτυχές που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και νομίζω ότι το ψήφισμα αυτό αναφέρει όλες τις πτυχές λίγο πολύ που πρέπει να λάβουμε υπόψη από την αναπτυξιακή σκοπιά. Δύο πράγματα ε, θεωρούμε πολύ σημαντικά. Από τη μία, να εξασφαλιστεί ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες μπορούν να συμμετέχουν επίσης όρις στην, ε, στο διεθνές θεματολόγιο τη φορολογική διακυβέρνηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδίω ό,τι αφορά ε, τη διάβρωση της βάση και αντιμετώπιση των κερδών. Η ομάδα των 20 κυρίω καθόριζε το θεματολόγιο. Τώρα όμως θέλουμε να έχουμε ένα πλαίσιο αλληλέγγυο συμπερίληψη όλων, inclusive framework, δηλαδή όλες οι χώρες να συμμετέχουν στην διαδικασία BEPS και στη διαδικασία διακυβέρνηση, ε, την καθορισμό προτίμων και κανόνων, Επίση όλε όπω είπα. Μέσω του όσα επεξεργαζόμαστε, επεξεργαζόμαστε μια συμφωνία, ένα σύμφωνο, ώστε να παράσχουμε τεχνική χρηματοοικονομική βοήθεια στι χώρε αυτέ για να συμμετάσχουν στη διαδικασία διακυβέρνηση. Αυτή είναι μια πτυχή. Εξίσου σημαντικό για μα. είναι και ο ρόλο των ΗΠΑ στο πλαίσιο τη Διεθνού Φορολογική Διακυβέρνηση. Στηρίζουμε μέσω συνεργασίας με τη Φορική Επιτροπή το έργο των υποεπιτροπών τη Φορική Επιτροπή των ΗΠΑ, με τη συμμετοχή ιδίω των ανεψωμένων χωρών που επιτροπέ, ώστε να μπορούν να φέρουν σε πέρα το έργο του. Ε, και τώρα θα δημιουργήσουμε μία ακόμα σύμβαση με τα Ηνωμένα Έθνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να ενισχύσει το έργο τη Φορική Επιτροπή του ΟΗ. Αυτές είναι οι δύο πτυχές που ήθελα να αναφέρω, που είναι συγκεκριμένε δράσει που θα χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε οι χώρε να μπορούν πραγματικά να συμμετέχουν περισσότερο σε αυτή την παγκόσμια διαδικασία φορολογική διακυβέρνηση. Δεν είναι να σταματάμε εδώ όμω. Θα πρέπει αυτό το domestic revenue mobilization να στηριχθεί και με συγκεκριμένε πράξει, ε, δράσει ε, για την ανάπτυξη υποδομών, δημιουργία ικανοτήτων Θέλουμε την προσέγγιση των καλύτερων δαπανών. Και πρέπει να στηρίξουμε τις προσπάθειες ε, των χωρών, εταίρων, για να αυξηθεί η κινητοποίηση αυτή, αλλά και κατά τρόπο που θα αντιμετωπίζει και τα προβλήματα ανισότητας. Δεν θα αυξάνει μόνο τους τελεστές, και έχουμε για αυτό το σκοπό παγκόσμια, περιφερειακά και εθνικά προγράμματα. Σε παγκόσμιο επίπεδο συνεργαζόμαστε με πολλούς εταίρους. Πάντοτε, όχι μόνο με στόχο, αλλά με γνώμονα τη συνεργασία μας με τους χώρες εταίρους επιτόπου, για να βελτιώσουμε και να παράσχουμε βοήθεια στις μεταρρυθμιστικές πολιτικές, φορολογικής ε, Συνεργαζόμαστε με Παγκόσμια Τράπεζα, Βαλτάνη ΤΑΦ, τον ΟΗΕ και με τον ΟΣΑ συνεργαζόμαστε για να βοηθήσουμε με παγκόσμιε πρωτοβουλίε τι ε, ανεψόμενε χώρε να βελτιώσουν την κινητοποίηση των εγχώριων φορολογικών εσόδων. Επίση, έχουμε ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα μέσω της Παναφρικανικής Χρηματοδότησης. Έχουμε συνεργασία με τέσσερις. ΑΤΑΦ, Άφρασα και άλλους δύο φορείς μια ιδιαίτερη ε, συνεργασία μας ενός προγράμματος, το οποίο νομίζω ότι απτά δείχνει πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις χώρες οποίες Σαχάρα στην προκειμένη περίπτωση να φέρουν σε πέρα, τις, σε πέρα σε τη, τα μέτρα του θεματολογίου για την κινητοποίηση εγχώρων φορολογικών εισόδων. Διάσκεψη κορυφής Αφρικής Ένωση Αφρική. Εκεί συζητήθηκε αλλά δεν θέλω να υπερβώ το αρμοδιότητέ μου και να πω πολλά από αυτό, αλλά μπορώ να πω απλά ότι συζητήθηκε το θέμα των παράνομων οικονομικών ορών και η συνέχεια που θα πρέπει να δοθεί στην έκθεση Ιμπέκη τη παρανοχων οικονομικέ ώρε από την Αφρική. Είπαμε ότι πρέπει να είναι και αυτό ένα θέμα θα μπορούσε να προταθεί να συμπεριληφθεί στο θεματολόγιο και εκεί σταματώ, δεν μπορώ να υπερβώ τι αρμοδιότητέ μου, παραλαμβάνω. Το θέμα είναι ο πολιτικό διάλογο μεταξύ των διαφορών εταίρων για να αντιμετωπιστεί αυτό το πολύπλοκο ζήτημα. Αυτό θέλουμε. Και σε επίπεδο αναπτυξιακή συνεργασία, αυτό που μπορούμε να κάνουμε και που μπορούμε να βοηθήσουμε, γιατί είπα, έχουμε αυτή τη μεταρρυθμιστική ατζέντα. Έχουμε προγράμματα. Και κάτι άλλο τελευταίο και σημαντικό είναι σε εθνικό επίπεδο, πως ξέρετε. Συχνά παρέχουμε δημοσιονομική ενίσχυση στην αναπτυξιακή συνεργασία. Θα εστιάσουμε πολύ περισσότερο στις στα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης που θα θέλουμε να τα συνδυάσουμε με τα μέτρα μας για την κινητοποίηση εγχώριων φορολογικών εσόδων για να μπορεί να υποστηριχθεί αυτή η δεύτερη διαδικασία πιο πολύ μέσω και της δημοσιονομικής ενίσχυσης όπου αυτό ε, είναι σκόπιμο. Αυτά μπορούμε να κάνουμε από την και σκοπιά. Είπα βέβαια ότι σε καμία περίπτωση δεν εξαντλούμε εκεί τι προσπάθειες για την καταπολέμηση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών. Αν μου επιτρέπετε τώρα, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον συνάδελφό μου από τη Δέλτα ΤΖΑΣΤ, ο οποίο θα σα μιλήσει για το ξέπλυμα του χρήματο και για του πραγματικού δικαιούχου. Ευχαριστώ. Thank ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Λέγομαι Τόμας Γιόγκριστ από την ε, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης ε, και Καταναλωτών από τη μονάδα του οικονομικού εγκλήματος και ασχολούμαστε με την καταπολέμηση της ε, νομιμοποίησης ε, παράνομων εσόδων. Εργαζόμαστε πάνω σε ένα ψήφισμα που περιγράφει τα πιο σοβαρά προβλήματα που επηρεάζουν τις χώρες ΑΚΕ. Η νομιμοποίηση παράνομων εσόδων και η χρηματοδότηση ε, για τρομοκρατικές ενέργειες αποτελούν σημαντικά προβλήματα για την περιοχή αυτή. Είναι όμως και παγκόσμια προβλήματα και αυτό σημαντικό είναι να αναζητήσουμε διεθνείς λύσεις. Η αποτελεσματική διεθνή συνεργασία στον τομέα αυτών είναι απαραίτητη. Καλούμε λοιπόν τις χώρες ΑΚΕ να διασφαλίσουν την πλήρη και προσεκτική εφαρμογή των συστάσεων της ειδική ομάδας, της Task Force και να δημιουργήσουμε στεναρά προληπτικά συστήματα για να μπορέσουν να καταπολεμήσουν αυτά τα επικίνδυνα φαινόμενα εκ των έσω. Όσον αφορά το πολύ σημαντικό θέμα της οικειοποίησης, επικροτούμε τη συμπερίληψη της σχετικής παραγράφου στο ψήφισμα. Ο τύπος ιδιοκτησίας ε, των ε, εταιριών και άλλων φορέων καθώς ε, και όλων των νομικών σχηματισμών όπως είναι τα καταπιστευματικά ταμεία θα πρέπει η ιδιοκτησία όλων αυτών να δημοσιεύεται σε συμμόρφωση με όλους τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων το ε, πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όσον αφορά την πραγματική κυριότητα είναι πολύ ε, σημαντικό θέμα και ξεπερνάει τα όσα γίνονται σε άλλες δικαιοδοσίες επάνω στο θέμα αυτό. Σας παραπέμπω και πάλι στις συστάσεις σχετικά με, την, με τους πραγματικούς δικαιούχους. Θέλουμε λοιπόν τώρα ε, να δημιουργήσουμε περαιτέρω αναλυτικούς κανόνες ε, και μπορούμε να παράσχουμε περαιτέρω ευηρογνωσία πάνω στο θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συνέπεια προωθεί ε, διεθνή πρότυπα για τους ε, πραγματικούς δικαιούχους καθώς ε, και για την αποτελεσματική εφαρμογή και στο πλαίσιο της ειδική ομάδας ε, για την σχετική δράση και στο πλαίσιο των G20. Είναι απαραίτητο οι σχετικές συστάσεις να είναι πλήρεις και να εφαρμοστούν με συνέπεια από όλε τι δικαιοδοσίε για να αποφύγουμε τα παραθυράκια. Διότι, όπως ε, σας είπα, το θέμα της νομοποίησης παράνομων εσόδων και της ε, ε, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι παγκόσμια προβλήματα τα οποία πρέπει να λύσουμε από κοινού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επρόκειτο να μιλήσει και κάποιος ποιο τρίτο άτομο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καταφτάσει ακόμα. Ναι, πράγματι, ένα συνάδελφο από τη Γενική Διεύθυνση ε, Φορολογία ε, πρόκειτο να καταφτάσει. Ωραία, θα δώσουμε το λόγο στους ευρωβουλευτές ε, και εάν καταφτάσει στο μεταξύ ο συνάδελφός σας θα μπορέσει να κάνει κάποιες... θα μπορέσει να παρουσιάσει τις παρατηρήσεις του. Θα θυμάστε ότι στη χθεσινή συνάντηση αναφέρθηκαν θέματα που είχαν θυχθεί από τα νησιά παρβάτος Μπορούμε να ακούσουμε διάφορες παρατηρήσεις. Ε, ο Μαυρίκιος έχει το λόγο, Χίνδια Συγγνώμη, δεν φοράω τα γυαλιά μου. Ο Μαυρίκιος, Νιγηρία. Τρινιντάτ και τον Μπέικο and uh, I I see um, South Africa and Barbados. Yes? Barbados will come after, if you don't know. Okay. Thank you, Chair. Yes. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίασή της. Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ στην παράγραφο 20 του ψηφίσματος ε, του και αυτά που συνέβησαν ε, τον Δεκέμβριο του 2016 στην Κένια και να κάνω τις ε, εξής παρατηρήσεις. Καταλαβαίνουμε ότι το σκεπτικό των δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής ε, είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι εναρμονισμένη η φοροαποφυγή σε όλη την Ήπειρο. Έτσι λοιπόν, όπω και σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν υπάρχουν ε, συνθήκες ίσου ανταγωνισμού σε θέματα φορολογίας. Επίσης, καταλαβαίνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την πρότασή τη ε, για μια κοινή φορολογική βάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, CCTB. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή η κοινή φορολογική βάση δεν θα εξαλείψει από μόνη τη ε, ε, τον επιβλαβή φορολογικό ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθότι τα κράτη-μέλη θα συνεχίσουν να είναι ελεύθερα να επιλέξουν μείωση ε, της εταιρική φορολογικής βάσης. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει διεθνής ή ευρωπαϊκός κοινός κατάλογος, ο κοινό κατάλογος ε, θα επιφέρει διακρίσεις και θα είναι αυθαίρετο ε, και θα οδηγεί σε μονομερή μέτρα. Επικροτούμε Μάλλον ε, επικρίνουμε την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμπεριλάβει χώρες όπως είναι ο όπου έχει εφαρμόσει σωστά όλα τα πρότυπα. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί οι χώρες μας έχουν αποτελέσει αδίκως στόχο. Και για όλους τους λόγους αυτούς η αντιπροσωπεία μου ε, είναι δυσαρεστημένη που δεν υπάρχει διάλογος με την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τον κατάλογο αυτών, διότι δεν πιστεύουμε ότι είναι δίκαιος ο κατάλογος αυτός και είναι εις βάρος της εταιρικής μας σχέσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, η γυρία. Ευχαριστούμε κυρία Συμπρόεδρε. Όπως και ο συνάδελφος από τον Μαυρίκιο, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μίλησε για αυτό το σημαντικό θέμα. Όπως συμβαίνει πάντα όμως, ερχόμαστε, ακούμε, ψηφίζουμε ψηφίσματα και όταν ακούμε τι δράσεις αναλήφθηκαν μετά από τα ψηφίσματα αυτά, διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε φτάσει πουθενά. Ακούμε αυτά που έχουμε να ακούσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά εγώ δεν έχω την αίσθηση ότι κατάλαβα κάτι για δράσεις, συγκεκριμένες δράσεις που να αναλαμβάνονται προκειμένου να πετύχουμε τόσο αναφέρονται στο ψηφισμό μας. Για παράδειγμα, υπάρχει το θέμα της νομοποίησης παράνομου χρήματος και η χρηματοδότηση τρομοκρατίας κλπ. Επ' αυτού δεν φτάνει να πούμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε με περιορισμούς και πώς θα συνεισφέρουμε σε αυτό, εφόσον το στερνιστούμε. Οι αφρικανικές χώρες, όταν συζητήθηκε αυτό το θέμα, είπαν ότι πόροι κάποιων αφρικανικών χωρών έχουν τύχη κατάχρησης από κάποιους πολιτικούς και που παράνομα κατάφεραν να πάρουν στα χέρια τους τεράστια χρηματικά ποσά που φτάσανε σε χρηματοοικονομικούς παραδείσους στην Ευρώπη. Ποια είναι η σχέση λοιπόν των χωρών αυτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα που σας μιλάω, αναφέρομαι στην Ιγυρία συγκεκριμένα. Τα πετροδόλαρα πηγαίνουν στις ελβετικές τράπεζες. Εντοπίστηκαν ως παράνομη χρηματοοικονομική ροή. Πήγαν τα θέματα αυτά στα δικαστήρια στην Ευρώπη, αλλά δεν έχουμε την βοήθεια που περιμέναμε ότι θα είχαμε. Περιμέναμε κάτι συγκεκριμένο σαν βοήθεια από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει των όσων αναφέρει το ψηφισμά μας. Δυστυχώς όμως Έτσι λοιπόν έχουμε διαπιστώσει ότι χρήματα πέρασαν παράνομα, αποδείχθηκε σε πολλές περιπτώσεις ότι ήταν παράνομο χρήμα Οπότε, τι περιμένετε να αποτελέσει αποτρεπτική δράση. Πώς θα γίνει αυτή η αποτροπή για άλλους που θα θέλανε να κάνουν το ίδιο αν δεν διαπιστώσουν ότι όντως αποτρεπτικά μέτρα λειτουργούν. Λοιπόν, να προσπαθήσουμε να είμαστε σύντομοι, παρακαλώ, για να μπορέσουν όλοι να πάρουν το λόγο. Παρακαλώ. Σε μένα το λέτε συγκεκριμένα. Ευχαριστώ. Πάντως ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία αυτή να μιλήσω εκ μέρους της χώρας μου, Τρινιδάδ και τον Πάγκο. Που προσπαθεί με συμμετοχή της σε πρόγραμμα να συμμετάσχει στο Διεθνές Φόρουμ για τη Διαφάνεια με ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά φορολογικά ζητήματα. Είχαμε την ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλάει για τους φορολογικούς περιορισμούς, κάτι το οποίο έχει προσέξει η χώρα μου και προχωράει σε ρυθμιστικές υποχρεώσεις, έτσι όπως προβλέπονται από το φόρουμ του ΟΣΑ. Μεταξύ άλλων, η χώρα μου, Τρινιτάδα και το Μπάγκο, θέλει διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελέσματα, δεδομένου ότι δεν θέλουμε να χάνονται πόροι από τους λίγους που έχουμε μέσα σε τέτοιες ροές παράνομες. Οπότε θέλουμε διευκρινήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις περιπτώσεις που διαπιστώνονται αποκλήσεις ανάμεσα στις προδιαγραφές που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και εκείνες που προβλέπει το φόρουμ του ΟΣΑ. Και που τελικά ε, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση απόλυτη με τις ε, αποφάσεις του ΟΣΑ. Εμείς θέλουμε να υπάρχει συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του φόρουμ του ΟΣΑ. Εμείς επιστήμουμε την προσοχή σας στην παράγραφο 14, η οποία τι λέει, λέει ότι ζητάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει περισσότερο ενεργό ρόλο προκειμένου να προσφέρει χρηματοοικονομική αρρωγή για να συμμορφωθούν οι χώρες προς τη διατάξη εκείνες οι οποίες βοηθούν να υπάρξει συμμόρφωση προς τις διατάξεις καταπολέμησης παράνομων χρηματοοικονομικών ορών. Η Τρινιδάδη και το Πάγκο λοιπόν θέλει να προτείνει διάταξη με αρρωγή προς τις αναψώμενες χώρες για να αναπτύξουν την ικανότητά τους να συμμετάσχουν σε αυτόν τον πρόσφατα προτινόμενο διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να εφαρμοστούν οι προδιαγραφές που προβλέπει το Φόρουμ το ΣΑ. Εάν υπάρξει αρρωγή αυτή, η Τρινιδάδη και το Πάκο θέλει να προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να καθορίσει χρονοδιάγραμμα και να διευκολύνει την εφαρμογή των ε, προδιαγραφών του ΩΣΑ με αρρωγή, έτσι ώστε να μπορούν και αυτές να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόεδρος, σε ευχαριστούμε. Νήσι ε, Κομόρες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να συμφωνήσω με τα όσα είπε ο εκπρόσωπος της Γουινέα και τα όσα είπε ο εκπρόσωπος της Νιγηρίας. Θα ήθελα να γνωρίζω, γιατί κατά τη διάρκεια τη συζήτηση για το ψήφισμα αυτό, είχαμε μιλήσει για την ε, διεύρυνση ε, για παράνομες δραστηριότητες ε, όπως ε, το εμπόριο ναρκωτικών και η πορνεία. Μια πρακτική για ξέπλυμα χρήματος, το οποίο καταλήγει συνήθως σε ε, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε ευρωπαϊκό έδαφος. Πρέπει να μιλήσουμε λοιπόν για τρομοκρατία, χρηματοδότηση αυτής κτλ. Πρέπει να μιλήσουμε για κάτι πρακτικό, γιατί πρόκειται για συγκεκριμένες χώρες και για αγαθά που, και για χώρες που ζητούν ευρωπαϊκή βοήθεια, ενώ έχουν τα μέσα. Τι κάνετε σήμερα, ποια είναι η λύση και ποια είναι η αντίδρασή σας ε, συγκεκριμένα. Οι χώρες ΑΚΕ και κυρίως οι αφρικανικές χώρες έχουν λαιλατηθεί, όχι από σας, ίσως από ορισμένου άνδρες και γυναίκες των χωρών των ίδιων. Πρόκειται για αγαθά τα οποία έχουν ε, αποκτηθεί με λάθος τρόπο. Εσείς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι κάνετε για να αντιμετωπίσετε τα αγαθά αυτά που βρίσκονται σε ευρωπαϊκό έδαφος. Πριν να μιλήσουμε για τα χρήματα της τρομοκρατίας, πριν να μιλήσουμε για βοήθεια και ρογή, είμαστε εδώ οι χώρες ΑΚΕ να λύσουμε το πρόβλημα μιας και διαπαντός, γιατί εμείς ε, ε, διαρκώς ε, είμαστε σε αυτή την... Ε, διαρκώς πίσω. Μας ξεπερνάτε. Πρέπει να, πρέπει εγκαταλείψουμε αυτό που μου αρχίσαμε να κάνουμε για να ακολουθήσουμε το ρυθμό. Ποτέ δεν λύνεται ένα πρόβλημα. Πηδάμε στο επόμενο. Και εγώ θα ήθελα να μπορέσουμε να δώσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Και οι απαντήσεις αυτές πρέπει επιτέλους να δοθούν. Εντάξει, Νότιος Αφρική και σας παρακαλώ να είστε σύντομος. Μάλιστα, Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Εγώ θέλω να στηρίξω τα όσα είπε ο δελφός μου για την διάσκεψη κορυφής Αφρικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό το θέμα θα είναι στα, στο θεματολόγιο τον Νοέμβριο. Και ακριβώς επειδή Αγαπητοί Πρόεδρε, 60 δις ετησίως φεύγουν από την Αφρική και αυτά τα μισά είναι από εμπορική δραστηριότητα καθαρά και τα άλλα μισά είναι από τις ε, ε κέρδη από ψεύτικες υπερτιμολογίες, υποτιμολογίες και ούτε καθεξές. Πάντως ε, θα πρέπει να πούμε ότι αυτά τα θέματα είναι ε, αλληλοσυνδεόμενα. Οποτεδήποτε δηλαδή συζητάμε παράνομη ε, ε, εκροή κεφαλαίων, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την παράνομη ροή, μάλλον τη ροή ε, χρημάτων ε, προς και από την Αφρική που είναι παρόνομη και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν μπορεί να διαφεύγουν επειδή αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο και ανήκουν σε πολυεθνικές εταιρείες ε, οι οποίες ε, τα μοιράζουν μεταξύ τους και το κάνουν ξανά ενθαρρύνοντας και πιέζοντας την οικονομία αναλόγως. αστάθεια, πίεση που, που, που οδηγεί αυτές τις πολυεθνικές στο να φύγουν από τις χώρες μας, γιατί αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο. No, before I said uh, Burundi and then St. Lucia and then Barbados. Burundi. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δίνετε ακόμη μια φορά το λόγο. Και εγώ έχω τις ίδιες εντυπώσεις όπως ο συνάδελφος από τις νήσους Κομόρες. Θα ήθελα να επιμείνω ακόμα μια φορά ότι οι ροές αυτές οι, οι χρηματοπιστωτικές που αφήνουν τις αφρικανικές χώρες ή τις χώρες ΑΚΕ προς τις ευρωπαϊκές χώρες θέλω να ρωτήσω τους ευρωπαίους ε, συναδέλφους τι κάνουν για να σταματήσουν αυτές τις ροές προς την Ευρώπη γιατί γνωρίζουμε ότι είναι ένας τρόπος λαϊλάτησης των αφρικανικών χωρών. Επίσης θέλω να επιμείνω για το μήπως δεν πρέπει αυτές να ποινικοποιηθούν οι ροές, δίνοντας το μήνυμα ότι κάθε χώρα που λαμβάνει αυτά τα χρήματα θα πρέπει να τα στέλνει πίσω στην χώρα προέλευσης. Θέλω να επιμείνω σε αυτό γιατί ξέρετε αν πιάσουν τους ε, εγκληματίες ή τους μετανάστες υπάρχει τρόπος να τους επιστρέψουν στη χώρα προέλευσή του. Τα χρήματα γιατί δεν τα επιστρέφουν, στη χώρα προέλευσή τους. That's a good, that's a good one. Καλή ερώτηση. λοιπόν, για γελουκία. Difficult to send than, than human beings, eh? Είναι πιο δύσκολο να στέλνει καλής χρήματα. Κυρία Πρόεδρε, Μια διευκρίνηση θα ήθελα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μίλησε για τους πραγματικούς δικαιούχους να δημοσιεύονται, να δημοσιοποιούνται. Σε ποιον όμως θα ήθελα να ξέρω. Θα μπορούσε να απαντήσει παρακαλώ. Εντός. παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Συμπρόεδρε που μου δίνετε τη δυνατότητα και πάλι να πάρω το λόγο πάνω στο θέμα του αντικτύπου των παράνομων ε, χρηματοοικονομικών ροών. Ε, τα νησιά Παρβέιτος συμφωνούν ε, ότι η καταπολέμηση αυτού του προβλήματος είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ακεραιότητας του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος. Δεν είναι όμως όλες οι χρηματικές ροές παράνομες. Η διάκριση θα πρέπει να γίνεται ανάμεσα σε αυτό που αυτή τη στιγμή ορίζεται ως παράνομη ε, χρηματική ροή και άλλες κατηγορίες ε, που λάθος θεωρούνται τέτοιες, ώστε ε, να μην καλύπτονται χώρες αδίκως. Εν τα νησιά Παρπέιτος ε, έχουν υπερασπιστεί τον τομέα τους, ε, τον χρηματοοικονομικό τομέα που υπάρχει εδώ και 20 χρόνια. Αλλά μας ε, κατηγορούσαν ήδη τότε σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη, αλλά έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ο ΣΑΑ τώρα θεωρεί ότι στην Καραϊβική ε, τα χρηματοοικονομικά συστήματα γενικά συμμορφώνονται με τους κανόνες ε, σχετικά με την ε, συνεργασία σε φορολογικά θέματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εταίρος τον ε, παρπείτος και ο ΣΑ είναι το θεμητό όργανο για ε, τον καθορισμό των προτύπων ε, για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών. Και τα νησιά Παρπείτος θέλουν να συμμετέχουν ενεργά, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση αγνοεί τις αποφάσεις αυτού του φορέα και ακολουθεί το δικό της δρόμο. Το θέμα λοιπόν αυτό δημιουργεί προβλήματα για τα νησιά Παρπέιτος διότι η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή ε, συνδέονται κάθε φορά, ενώ η μία πρακτική είναι παράνομη και η άλλη είναι νόμιμη. Και βλέπουμε να επαναλαμβάνεται αυτό στην διατύπωση της διακήρυξης ε, του Ναϊρόμπι, της Περσινής. Επίσης, ε, τα Περπέιτος αναγνωρίζουν ότι η σύγχυση των δύο αυτών θεμάτων έχει γίνει πια ευρέως ε, αποδεκτή σε πολλά κείμενα. Αυτό όμως είναι ανεύθυνο. Υπάρχουν μηχανισμοί διασφάλισης για την εξέταση οποιασδήποτε επιχείρησης δημιουργήσει υπεράκτια εγκατάσταση στα νησιά Μπαρπέιτο και γίνονται έλεγχοι σχετικά με την ε, καλή πίστη των εταιριών αυτών ε, σε συνεργασία με αναπτυγμένες χώρες. Δεν είναι κάτι αυτό που κάνουμε μόνοι μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε άδικη πρακτική μαύρης λίστας ε, τον Ιούνιο του 2015 με δημοσίευση ε, δικαιοδοσιών ε, που δεν συμμορφώνονται χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τις χώρες αυτές. Και δυστυχώς φαίνεται να υπάρχει αυξανόμενη τάση για λήψη μονομερών αποφάσεων όσον αφορά το πώς θα πρέπει να χειριζόμαστε θέματα φορολογίας και διακυβέρνησης και η κατάσταση επιδεινώθηκε με την ε, δημιουργία πίνακα αποτελεσμάτων ε, όπου αναφέρονταν ε, ο βαθμός συμμόρφωσης με βάση τρία κριτήρια, τη διαφάνεια, την ανταλλαγή πληροφοριών και τον φορολογικό ανταγωνισμό. Αμφισβητείται ο φορολογικό συντελεστή που εφαρμόζεται από τι χώρε αυτέ και η ηρωνία εδώ είναι ότι εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει συμφωνία ε, για κοινή φορολογική βάση ε, με τρίτες χώρες. Κυρία Πρόεδρε, μετά ξεκίνησε η διαδικασία ελέγχου, screening, και ζητήθηκαν πληροφορίες από τις πρωτεύουσες σχετικά με άτομα ε, που εμπλέκονταν σε διάφορες φορολογικές υποθέσεις. Τα νησιά Μπαρμπέιτος συμμορφώθηκαν με το αίτημα αυτό. Το άρθρο 12 της σχετικής συμφωνίας προβλέπει διαβουλεύσεις ε, μεταξύ των μερών εάν υπάρχει κάποιο θέμα που να επηρεάζει τη σχέση μεταξύ των χωρών αυτών. Ε, κατά την ε, συνάντηση πρέσβεων του Μαρτίου του 2017 η ευρωπαϊκή πλευρά δήλωσε σαφώς ότι δεν θα ξεκινήσει διαβουλεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 12 με τις χώρες ΑΚΕ για το θέμα αυτό. Αυτό είναι ατυχές. διότι ε, αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σημαντικές επιπτώσεις ε, για κάποιες χώρες όσον αφορά το εμπόριο και τις υπηρεσίες που παρέχουν. Και σας καλούμε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή. Ελπίζουμε ότι έτσι θα αληθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες ε, των χωρών που εμπλέκονται. Θα ήθελα να τονίσω ότι όλα αυτά αντίκυνται στο πνεύμα του Κοτονού. Όπως είπα στον Ναϊρόμπι και επαναλαμβάνω εδώ πέρα, τα νησιά Παρβέιτος, όπως και οι περισσότερες ε, οικονομίες της Καραϊβικής ε, βασίζεται στις υπηρεσίες. Έχουν πολύ στενό ε, δημοσιονομικό περιθώριο. Και ο υπεράκτιος τομέα μαζί με τον τουρισμό αποτελούν την, την βασική πηγή της οικονομίας μας. Και δεν ε, έχουν ε, καταβληθεί προσπάθειες ε, για να γίνει κατανοητή η κατάσταση χωρών όπως είναι τα νησιά Μπαρμπέιτος. Η ζημιά στους τομείς της υπεράκτησης οικονομίας και του τουρισμού δεν έχουν γίνει κατανοητές. Είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε σωστά τι εννοούμε όταν μιλάμε για παράνομες οικονομικές ροές, ε, όχι απλά να κάνουμε γενικεύσεις ε, που να θεωρούμε ότι ισχύουν για όλες τις χώρες. Θέλουμε λοιπόν να δώσουμε τέλο στι παράνομε οικονομικέ ροέ ε, και να φροντίσουμε να ξεχωρίσουμε την ήρα από το στάρι. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, Περπέιτο. Νομίζω ότι αυτό ήταν απαραίτητο, διότι τέθηκαν πολλέ ερωτήσει χθε. Σα ευχαριστώ πολύ που κάνατε την σχετική διευκρίνηση. Προτού να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι μπορώ και εγώ να κάνω μια ερώτηση. Παράγραφος Β. Στο έγγραφό μας. Αναφέρεται σαφώς ότι οι παράνομες χρηματοοικονομικές ροές έρχονται από τρεις τομείς. Φοροαποφυγή, πλαστογράφηση πιστοποιητικών καταχρηστική, ε, καταχρηστικές τιμές μεταβίβασης και εγκληματικέ δραστηριότητε, όπως είναι η εμπορία ανθρώπων, ε, η διακίνηση ναρκωτικών κλπ. Το δικό μου ερώτημα λοιπόν είναι τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις τιμές μεταβίβασης ε, και την ψευδή ταμολόγηση από τις ε, πολυεθνικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την έκθεση, αυτές οι πρακτικές συμβάλλουν κατά τα δύο τρίτα στις ε, παράνομες μετα... Ε, οικονομικές ροές από τις χώρες μας. Θα σας παρακαλούσα να απαντήσετε όσο γίνεται πιο γρήγορα, διότι μας μένει λιγότερο από μισή ώρα. Ακριβώς στις 7 θα σταματήσει η διερμηνία και έχουμε ακόμα ένα θέμα, τη γαλάζια οικονομία στην ημερήσια διάταξη. Σας παρακαλώ λοιπόν να είσαστε όσο γίνεται πιο σύντομη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα δώσω μετά το λόγο στον συνάδελφό μου από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας που θα απαντήσει σε μια ευρία γκάμα ερωτήσεων ε, που είχαν όλες την ίδια κατεύθυνση. Αναφέρομαι στο θέμα που έθιξαν ο Μαυρίκιος, ε, το Trinidad και το Μπέικο, καθώς και τα νησιά Μπαρμπέιντος. όσον αφορά την ε, τεχνική υποστήριξη και την οικοδόμηση δυναμικού στον τομέα αυτών. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές, ε, είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο πάνω στο θέμα αυτό. Και η γενική μας ε, διεύθυνση για την διεθνή αναπτυξιακή βοήθεια έχει σχετική εντολή και ευχαρίστως ε, να έρθει σε επαφή ο αρμόδιος ξεμοτούχος της χώρας σας με την πρεσβεία μας ε, στη χώρα σας για να συζητήσουν το θέμα αυτό και να φροντίσουν να παρασχεθεί τεχνική βοήθεια στον τομέα αυτόν. Είναι πολύ σημαντικό τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης και το θέμα αυτό δεν ε, συνδέεται αποκλειστικά με την δημοσιονομική στήριξη. Υπάρχουν ε, ταμεία βοήθειας για το θέμα αυτό. Είναι λοιπόν μια προσφορά που μπορούμε να σας κάνουμε για να δείτε ότι είμαστε σοβαροί όσον αφορά την ρηξαγωγή διαλόγου και να ε, συνομιλήσουμε επικοδομητικά για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Όσον αφορά το θέμα που έθιξε η Πρόεδρος σχετικά με το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των τιμών μεταβίβασης και των παράνομων ε, χρηματικών ροών ε, στις πολυεθνικές. Όπως σας ανέφερα, το πρόγραμμα BEPS ε, του ΟΣΑ, το οποίο όμως τώρα έχει επεκταθεί με το πλαίσιο ώστε όλες οι χώρες που θέλουν να εφαρμόσουν το σύστημα αυτό για τη διάβρωση της φορολογικής βάσης ε, και τη μετέβαση των κερδών ε, μπορεί να το κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στόχο να ασχοληθεί με θέματα BEPS και, και τιμών μεταβίβασης για να κλείσουν τα παραθυράκια και να περιοριστούν οι δυνατότητες των πολυεθνικών να ακολουθούν πρακτικές ώστε να ελαχιστοποιείται η φορολογία εκεί όπου επιτυγχάνεται η προσθέμενη αξία και όπου θα έπρεπε να πληρώνεται ε, εταιρικό φόρος. Στις μελέτες μας ε, για τις τιμές μεταβίβασης, ε, όπως έχουμε κάνει στην Δυτική Αφρική, συμπεριλαμβάνονται τα μέτρα του ασφαλούς λιμένα, Safe Harbor Measures, όπου εξετάζεται η δυνατότητα των χωρών της Δυτικής Αφρικής ε, να εφαρμόσουν καθεστώτα ώστε να μπορέσουν ε, να φρενάρουν αυτές τις πρακτικές από πλευράς των πολιεθνικών. Με το Διοικητικό Φόρουμ, ε, λοιπόν, στόχος είναι όχι μόνο να αντιμετωπιστούν τα εγχώρια θέματα δυναμικού, αλλά να αντιμετωπιστεί και η διεθνή πτυχή. Αυτό ήταν ένα παράδειγμα που ήθελα να σας δώσω. Θα δώσω όμως το λόγο στον συνάδελφο από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας που θα απαντήσει σε άλλες παρατηρήσεις που έγιναν. Ευχαριστώ πολύ. Really, um, um, I just Just a minute each, please. We are really running out of time. Ένα λεπτό παρακαλώ καθένας γιατί δεν έχουμε χρόνο. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, οι υπόλοιποι ενδεχομένω ε, θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή μαζί σας. Ένα λεπτό καθένας παρακαλώ. Οι εκπρόσωποι της Κομισιόν δηλαδή έχουν ένα λεπτό καθένας. Εγώ θα είμαι πολύ σύντομος. Νομίζω ο εκπρόσωπο από το Σάντα Λουτσία μίλησε για του πραγματικού δικαιούχου και σε ό,τι αφορά την οδηγία 2015-849 για τη χρήση συστημάτων. 5 Ιουνίου του 2015 δημοσιεύθηκε. Έλενα 4.1, σελίδα 73. Κεφάλαιο 3. Έχουμε εκεί τα στοιχεία ε, για τους πραγματικούς δικαιούχους. Άρθρα 30 για εταιρείε και λέει παράγραφος ότι τα κράτη-μέλη εξασφαλίζουν ε, ότι οι πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους είναι προσβάσιμες σε κάθε περίπτωση ε, ε, για τις αρμόδιες αρχές, μονάδες οικονομικών πληροφοριών χωρίς κανένα περιορισμό και τα λεγόμενα obliged entities, δηλαδή πιστοτικά, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και το καθεξής. Καθώς και οποιοδήποτε ιδιώτηση ή οργάνωση μπορεί να αποδείξει ότι έχει θεμητό ενδιαφέρον τα κράτη-μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους διατηρούνται σε ένα κεντρικό μητρό. Μπορεί να είναι εμπορικό μητρό ή κάτι άλλο. Το άρθρο 31 μιλά για τα καταπιστεύματα και εδώ μπορώ να σας πω μόνο ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουμε και ένα κεντρικό μητρό όταν έχει φορολογικές συνέπειες ε, η ύπαρξη ενός καταπιστωματικού ταμείου. Εν γέννη για τους πραγματικούς δικαιούχους είναι ένα θέμα που μπορεί να συζητηθεί στο πλαίσιο των διαφόρων φορέων της ΦΑΤΦ. πώς μπορεί να εφαρμοστεί δηλαδή. Και σε ό,τι αφορά για τις πληροφορίες. Έχουμε την ομάδα Έκμοντ για τις μονάδες των πληροφοριών που μπορεί να αξιοποιηθεί αυτή η ομάδα Έκμοντ για τη συλλογή πληροφοριών και βέβαια και μέσω της αμοιβαίας νομική συνδρομή. Αυτά έχω να πω προ το παρόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Θέλει κανεί άλλο το λόγο. Ένα λεπτό μόνο. Μόνο ένα λεπτό. Εσείς από την Κομισιόν ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομο και περιεκτικός. Αν άκουσα καλά ε, τις ανησυχίες, αυτές αφορούν κυρίως τη διαδικασία για το listing. Τι σχέση έχει με τη διαδικασία του ΩΣΑ, τη διαδικασία αυτή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ε, κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν το διάλογο ετέθησαν. Καταρχά, θέλω να πω ότι αν διαβάσετε το έγγραφο, το ψήφισμα, εκφράζει κάποιε ανησυχίε σε σχέση με τη αποφυγή, αναπτυξιακή, οντοδοκή οργανισμό κτλ. Νομίζω ότι αυτές οι ανησυχίες αντιμετωπίζονται, διασκεδάζονται μέσω του εγγράφου μας για την ε, διακυβέρνηση, που μιλάμε για διαφάνεια, ανταλλαγή πληροφοριών, δίκαιο ανταγωνισμό, και ΠΕΠΣ πρόσφατα. Αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωσης, νομίζω ότι ευθυγραμμίζεται σε μεγάλο βαθμό με τους στόχου του εγγράφου αυτού. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την πολιτική χρηστής φορολογικής πολιτικής, δεν άρχισε το 17 ούτε το 16. Είναι μια μακρόπνοη πολιτική που αναπτύσσεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ανακοίνωση Κομισιόν από το 2009 και με ειδική ανακοίνωση το 2010 έχουμε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια. Ο βασικός στόχος είναι να προωθήσουμε διεθνή φορολογικά πρότυπα προς τους εταίρους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω πρώτον της βοήθειας, αυτό κάνουμε εμεί και το είπαν και στην άρθρα πήγαμε τα ΔΕΦΚΟ, σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση εσωτερικών, συγγνώμη, εγχώριων φορολογικών εισόδων. Επίσης, και με άλλα μέσα που προωθούμε για την χρηστή φορολογική διακυβέρνηση. Σε ό,τι τα κριτήρια χρηστή φορολογική διακυβέρνηση, βασίζονταν για καιρό στην ανταλλαγή πληροφοριών. Το Global το Παγκόσμιο Φόρουμ είχε αναλάβει ε, το έργο αυτό. Τώρα έχει υπάρξει μια καιροποίηση και απόφαση του Συμβουλίου. Υπάρχει μια νέα συμφωνία μεταξύ και των 28 κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ποια θα πρέπει να είναι τα κριτήρια τη χρυσή φορολογική διεκπαίδευση, δηλαδή ανταλλαγή πληροφοριών, κατόπιν αιτήματο, αλλά και αυτόματη. Καλύπτεται επίση η αποφυγή επιζήμιων φορολογικών πρακτικών και τώρα συμπεριλήφθηκε η δέσμευση ε, να τηρούνται τα καθόλου τα πρότυπα δυνάμει του ΜΠΕΠΣΑ. Αυτό είναι θετικό. Δείχνει ότι η διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ε, πλήρως συμμορφούμενη με τα διεθνή τεκτενόμενα όπως από τον ΩΣΑ για παράδειγμα. Μπορεί να μην έχει προχωρήσει ίσως τόσο πολύ σε κάποιες πτυχές, όμως τα κριτήρια καταχώρησης που αποφασίζονται στο νοσιακό αποφασίζονται στο ε, διεθνές ε, έργο. Έρχομαι στο διάλογο. Και αν έχετε ερωτήσεις βεβαίως και ευχαριστώ να απαντήσω. Σε ό,τι αφορά το διάλογο. Αυτή η διαδικασία διαλογής, ε, καταχώρηση, το listing, screening, αναπτύσσεται από τα κράτη-μέλη και από το Συμβούλιο, γιατί από εκεί εκπηδάζει αυτή η διαδικασία και τρεις είναι οι φάσεις βασικά. Πίνακας αποτελεσμάτων, προκαταρκτική αναγνώριση και screening με εντατικό διάλογο αυτή τη στιγμή και τέλος το listing στα τέλη του χρόνου. που θα αποφασιστεί μετά το διάλογο και την ε, επιτυχή του έκβαση. Είναι σημαντικό λοιπόν οι χώρες που είναι σε επαφή με το Συμβούλιο να είναι σε επαφή με το Συμβούλιο για να παρουσιάσουν την περίπτωσή τους. Ε, ε νομίζω έληξε ο χρόνος μου. Αν θέλετε όμως να πάσω και σε άλλα ερωτήματα είμαι στη διάθεσή σας. Κοιτάξτε, πρέπει πραγματικά να σταματήσουμε τώρα. Οι δύο εισηγητέ, θέλετε να πείτε μια λέξη ο καθένα, οι δύο εισηγητέ. Και ο κύριο Στόλογεν, όχι. Really, Zambia, please allow us to, to, to move to the last topic because we will not have the advantage of having the, um, the interpreters uh, with us and this is a guest. So you want to go back to um, seven. Λοιπόν, ωραία, πάμε στο σημείο 7. Όπως γνωρίζετε, αλλάζει η οικονομία, ευκαιρίες και προκλήσεις για τις χώρες ΑΚΕ θα είναι το θέμα της επόμενης μας έκθεσης. Σήμερα επισήμως θα ορίσουμε τον ε, συνεισηγητές για αυτήν την έκθεση, μετά θα έχουμε μια δελαγή απόψεων. Ε, για αυτό το θέμα. Ενημερώθηκα ότι από την πλευρά ΑΚΕ ε, θα είναι ο κύριος Σαμούρη Μάντι Χασάνη και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι η κυρία Μαριέλ Ντεσαρνέζ, η συγγήτρια. Σα ευχαριστώ για την ε, αφοσίωσή του. Δυστυχώ η κυρία της Ανέ χρειάστηκε να φύγει λίγο νωρίτερα σήμερα και δεν θα μπορέσει σήμερα να σχολιάσει. Αλλά θα δώσω το λόγο στον κύριο Μάντι Χασάνη σε περίπτωση που επιθυμεί να κάνει κάποια προκαταρκτικά σχόλια γι' αυτό το θέμα. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η γαλάζια οικονομία προσφέρει στις χώρες εκεί την ε, δυνατότητα να ε, θεσπίσουν μια νέα πολιτική που θα βασίζεται στην... στον κοινωνικό τομέα. Τροφοδοτείται από τη φύση, συνδυάζει όλες τις οικονομικές δραστηριότητες που γίνονται στις ε, παραλίες, ε, στα, στις λίμνες, στα ποτάμια, στις θάλασσες, στο βυθό των ωκεανών, ε, και στους ε, ωκεανούς τους ίδιους. Αφορά όλες τις χώρες, ανεπτυγμένες και μη, και για τις χώρες ΑΚΕ. Το πρότυπο αυτό είναι η, πηγή ε, αιματηρών συγκρούσεων για αυτούς που τα έχουν. Γιατί η πράσινη οικονομία σημαίνει βαριές επενδύσεις που είναι απρόσιτες για τις περισσότερες χώρες. ΑΚΕ πέρα από τις επενδύσεις ε, πολλές φορές ε, συμβάλλει σε βλάβη, μάλλον ε, σημαίνει βλάβη για το περιβάλλον και γι' αυτό και η γαλάζια οικονομία για πολύ κόσμο παραμένει μια λύση αποτελεσματική όπου θα πρέπει όλοι να εγκύψουμε για να βρούμε λύσεις. Ελπίζω ότι για αυτή τη φορά δεν θα ζήσουμε την ίδια ιστορία και την ίδια φάση όπως για την κόκκινη οικονομία ε, και ότι αυτή η δαλασσιά οικονομία θα, θα συνεισφέρει στις οικονομίες όλων των χωρών όπου και να αυτές βρίσκονται και σε αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάντι. Να θυμίσω ότι για το χρονοδιάγραμμα ποιο είναι για τη σύνταξη της έκθεσης. Σήμερα είχαμε μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων. Τον Ιούνιο 2017 θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων επί τη βάση των εγγράφων εργασίας, οπότε μέχρι τον Ιούνιο θα υπάρχει το εγγράφο εργασίας. Τον Οκτώβριο φέτος εδώ στις Βρυξέλλες θα γίνει η παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης από τους συνεισηγητές και το Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους στην σύνοδο της ε, ΑΚΕ θα ε, εγκρίνουμε το σχέδιο ψηφίσματος. Τώρα θα κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων με τον David Carr που είναι ε, ειδικό για θέματα ναυτιλίας από την Μαλτέζικη Προεδρία η γαλάζια οικονομία είναι από τις βασικές προτεραιότητες της Μάλτα για το εξάμεινο της Προεδρίας της. Καθώς η Μάλτα βρέχεται από τα νερά, είναι ένα καλό παράδειγμα για να τονίσετε τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της γαλάζιας οικονομίας και σήμερα θα ακούσουμε πώς θα πρέπει οι χώρες εκεί να χρησιμοποιήσουν τις ευκαιρίες της γαλάζιας οικονομίας. Κύριε Κέρ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, καλησπέρα σε όλους και σας ευχαριστώ που μας καλέσατε την Προεδρία μας να σας περιγράψουμε ποιο είναι το πρόγραμμά μας σε σχέση με την γαλάζια οικονομία. Ε, όταν πρόκειται για την ευρωπαϊκή μπλε στρατηγική, γαλάζια στρατηγική, είναι μια στρατηγική που ξεκίνησε το 2012. Βέβαια, η γαλάζια οικονομία μας συνοδεύει εδώ και αιώνε, γιατί τα πλοία και τα καράβια εδώ και αιώνε ξεκίνησαν να πλέουν στα ευρωπαϊκά νερά. Όμως το 2012 η Κομισιόν ξεκίνησε μια διαδικασία μέσω της οποίας ε, ε, έκανε μια ανακοίνωση και ζήτησε από τα κατημέλη να κοιτάξουν προς τη θάλασσα και να δουν τι μπορούμε να έχουμε από τη θάλασσα όσον αφορά θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξης με βιώσιμο τρόπο. Τότε η Κομισιόν είχε τονίσει Πέντε κύριε τομεί, ανανεώσιμη ενέργεια, βιοτεχνολογία, παράκτια και θαλάσσιο, παράκτος και θαλάσσιος τουρισμός, ε, υδατοκαλλιέργειες και ε, θαλάσσιοι πόροι. Και ε, μετά από αυτή τη διαβούλευση ήρθε το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν να, να εξετάζουν και την ανάπτυξη μιας γαλάζιας στρατηγικής ώστε να εξασφαλίσουμε πως αυτοί οι πέντε τομείς προτεραιότητες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, ιδιαίτερα όσον αφορά τη βιωσιμότητα των τομέων αυτών. Βεβαίως, η στρατηγική ε, σημαίνει και την συνειδητοποίηση της καλής, της χρηστής διακυβέρνησης, ιδιαίτερα προωθώντας διεθνείς και τοπικές συμφωνίες, ιδιαίτερα την Αουγκλέους, μέσα στην οποία οφείλει να λειτουργεί η γαλάζια ε, οικονομία. Εφόσον υπάρχει νομική βεβαιότητα και χρηστή διακυβέρνηση, τότε εξελίσσεται ομαλά η διαδικασία. Στη διάρκεια λοιπόν της Προεδρίας μας εξετάσαμε αυτά τα πέντε έτη εξέλιξης της ευρωπαϊκής ε, μπλε οικονομίας, γαλάζιας οικονομίας και, και γαλάζιας στρατηγικής, ιδιαίτερα από την έναρξη της στρατηγικής αυτής υπήρξαν και πρωτοβουλίες όπως η ε, θαλάσσιος προγραμματισμός που δημιουργεί την νομική βεβαιότητα για τον σχεδιασμό ε, στα ευρωπαϊκά ύδατα. Τι κάναμε λοιπόν, κοιτάξαμε δύο πτυχές της γαλάζιας οικονομίας. Πρώτα απ' όλα είδαμε κοιτάξαμε να κάνουμε μια απογραφή του τι είχε γίνει τα τελευταία πέντε χρόνια και επίσης να δούμε τις περιβαλλοντικές ε, πτυχές των ωκεανών μας. Ε, όσον αφορά λοιπόν την ε, γαλάζια οικονομία, θέλουμε αυτή να προχωρήσει περισσότερο. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις όπως παράνομη αλληλεία, ή τα περιβαλλοντικά θέματα, τις κλιματικές αλλαγές, Θέλουμε λοιπόν η γαλάζια οικονομία να περάσει σε μια επόμενη φάση όπου πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες που γίνονται στους ωκεανούς να γίνονται με βιώσιμο τρόπο για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε, να προστατεύσουμε μάλλον τους ωκεανούς. Αυτό σε σχέση με την γαλάζια οικονομία όσον αφορά την απογραφή που κάναμε. Τώρα, επίσης εξετάζουμε διεθνώς τι σημαίνει διεθνής διακυβέρνηση των κενών. Όταν μιλάμε για μη ευρωπαϊκά κράτη, δηλαδή, πώς εξετάζουμε τους όρους συνεργασίας με χώρες εκτός Ένωσης. Έχουμε συζητήσει με κράτη της Μεσογείου που δεν ανήκουν στην Ένωση, για να ξεκινήσουμε αυτό που λέγεται Ε, στρατηγική της Μεσογείου, της λεκάνης της Μεσογείου, όπου με τρίτες χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο προσπαθούμε να καταρτήσουμε μια στρατηγική με βάση projects για να προωθήσουμε την ατζέντα της γαλάζιας ανάπτυξης εντός της Μεσογείου. Τώρα, όταν έχουμε να κάνουμε με την περιβαλλοντική πτυχή, όπως ανέφερα και προηγουμένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε μια νομοθεσία όσον αφορά την τον, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Επί τη βάση των οικοσυστημάτων γίνεται αυτό το πράγμα και δηλαδή βλέπουμε τώρα πώς χρησιμοποιούμε τους ωκεανούς και τις θάλασσές μας με βάση προσέγγιση ε, οικοσυστημάτων με οικοσυστήματα. Δηλαδή εξετάζουμε τα οικοσυστήματα όταν ε, ε, κάνουμε δραστηριότητες ή όταν σχεδιάζουμε, προγραμματίζουμε τις δράσεις μας για τις θάλασσες. Όλοι γνωρίζουμε τώρα την ατζέντα για το 2030 και ο στόχος είναι και υπάρχει και σε ένα ανακοινωθέν που πρόσφατα ε, εξέδωσε η Κομισιόν όσον αφορά τη διακυβέρνηση των ωκεανών και την ατζέντα για το μέλλον των ωκεανών μας Πήραμε λοιπόν αυτό το ανακοινωθέν και τον, στόχο βιώσιμο, τον βιώσιμο στόχο 14, υπαριθμών 14. Αυτή θα είναι η πρώτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου που υιοθετήθηκαν ε, και στα υπόλοιπα που είναι κοντά στην ε, οριστικοποίησή τους, ε, θεσπίσαμε πολιτική ατζέντα ώστε να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των ωκεανών μας και επίσης θα αναφερθούμε στη δυνατότητα ε, σχηματισμού δυνατοτήτων στα υπόλοιπα κράτη-μέλη και επίσης στη θέσπιση συνεργασιών με τρίτες χώρες. Φυσικά αυτά όλα η χρήση των ωκεανών και η ατζέντα της γαλάζιας ανάπτυξης δεν είναι σχετίζεται μόνο με την Ένωση. Έχει και μια διεθνή διάσταση όπου προφανώς ε, στατηγικά πλαίσια συνεργασίας με τρίτες χώρες ε, είναι πολύ σημαντικά για να εξασφαλιστεί η διατήρηση των ωκεανών και των θαλασσών μας. Επίσης κάτι που ενδιαφέρει αυτή την ομάδα έχει να κάνει με τη Διεθνή ε, Οργάνωση Ναυτιλίας, όπου εργαζόμαστε σε αγαστό πνεύμα συνεργασίας, ώστε να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή και την τήρηση των διεθνών συμφωνιών και μέσων. Η Μάλτα ως ε, θαλάσσιο κράτος και ως μέλος της Ένωσης αποδίδει μεγάλη σημασία στο ρόλο του Διεθνούς Οργανισμού ναυτιλίας όταν πρόκειται για την οικονομία για την, της γαλάζιας ανάπτυξης. Γιατί όπως ανέφερα χρειάζεται στεναρή και αποτελεσματική διακυβέρνηση. Βεβαίω έχουμε δει διάφορα θέματα σε αυτά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, όπως το θέμα των κλιματικών αλλαγών, το θέμα της ε, μη ρυθμιζόμενης ε, και παράνομης αλληλείας. Έχουμε θεσπίσει δεσμεύσεις όσον αφορά τα θαλάσσια απόβλητα που ξέρουμε ότι το 70% εξ αυτών προέρχονται από την γη. Και επίσης θέλουμε να προωθήσουμε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό αλλά και να εξασφαλίσουμε την προστασία των ωκεανών και των θαλασσών, γιατί αν, όλοι, αν οι θάλασσες και οι ωκεανοί δεν είναι υγιείς, δεν θα ανθίσει και η γαλάζια οικονομία. Να σας δώσω μια εικόνα τώρα του τι κάνουμε για τη γαλάζια οικονομία. Τα τελευταία πέντε χρόνια μετά την ευρωπαϊκή μπλε γαλάζια ε, οικονομία, πιστεύω πως θεσπίστηκε ένα σωστό πρόγραμμα, ένα υπόδειγμα που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν και άλλες ε, περιοχές ε, ώστε να εξασφαλιστεί ανάπτυξη και οι θέσεις απασχόλησης στις εν λόγω περιοχές. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση διερμηνής δέχτηκαν να ξεπεράσουν το χρόνο κατά 10 λεπτά. Να προχωρήσουμε μέχρι τις 7 και 10. Η Πρόεδρος ευχαριστεί ευγενικά του διερμηνείς για αυτό. Σας παρακαλώ όμως να εκμεταλλευτούμε καλά τον χρόνο αυτό. Υπάρχει κανείς που θέλει να πάρει το λόγο. Να θυμάστε ότι είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Ε, βλέπω τα νησιά Παρπέιτος. Υπάρχει κανείς άλλος. Παρπέιτος, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Sorry. The blue economy, like the green economy, η γαλάζια οικονομία όπως και η πράσινη έχει αρχίσει ε, να ε, λαμβάνει κεντρική θέση. Ε, τα Μπαρβέιτος όπως και άλλα μικρά νησιωτικά κράτη επικροτεί την εξέλιξη αυτή διότι η θάλασσα έχει άμεσο αντικτύπο στην ύπαρξή μας. Εμείς θα θέλαμε λοιπόν να δούμε αυτή τη νέα κατεύθυνση του θεματολογίου 2030 για βιώσιμη ανάπτυξη τους ε, στόχους 13 ε, και 14. Θα πρέπει να ε, γίνουν οι σύνδεσμοι με άλλα οριζόντια θέματα για να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών μας. Πρέπει να βρεθεί σωστή ισορροπία, να έχουμε καλύτερα μέτρα, να προστατεύσουμε τους ωκεανούς μας επίσης. Τα νησιά Παρμπέντος θεωρούν ότι αυτό αποτελεί κοινή ευθύνη συμπράξεων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Ε, οι ιστορίε επιτυχία σε τέτοιων συμπράξεων αποτελούν έναν τρόπο να προωθηθεί το θέμα αυτό. Υπάρχει κανείς άλλος που να θέλει να κάνει σχετική παρατήρηση, από ό,τι βλέπω όχι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να απαντήσει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Είμαστε ευγνώμονε που η Μαλτέζικη Προεδρία έχει δώσει προτεραιότητα στο θέμα αυτό και έχει οθετήσει αρκετέ από τι πρωτοβουλίε μα και τι προωθεί. Θα ήθελα να προσθέσω δύο ενημερωτικά θέματα, τα οποία ε, θα μας ενδιαφέρουν και σε σχέση με την έκθεση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει την εκπόνηση μελέτη σχετικά με ε, τη γαλάζια διάσταση στις πιο απόμακρες ε, περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιμένουμε να ολοκληρωθεί τον Μάιο. Όπως γνωρίζετε, οι πιο απόμακρες περιφέρειες βρίσκονται πολύ κοντά σε κάποιες από τις χώρες που εκπροσωπείτε εσείς και μπορεί να έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά και έτσι λοιπόν να υποφεληθούν και άλλες χώρες από τη μελέτη αυτή. Άλλη πρωτοβουλία που θα ξεκινήσει σύντομα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η πρωτοβουλία καθαρής ενέργειας για τα νησιά. Η καθαρή ενέργεια είναι φυσικά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τα πιο απομακρυσμένα νησιά που συχνά χρησιμοποιούν πολύ ε, ακριβές μορφές ενέργειας. Θα κλείσω εδώ. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Μαντή, παρακαλώ. Θέλετε να πείτε κάτι ακόμα, όχι, όχι δεν πειράζει. Mr. Kerr from Malta, you good? Okay. Well... Η Μάλτα, όχι. Α, ωραία. Καταφέραμε να ολοκληρώσουμε πριν τις 7 η ώρα. Ε, παρακαλώ χειροκροτήστε τους διερμηνείς, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Um, έτσι ολοκληρώσαμε τις σημερινές μας εργασίες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την εξαιρετική συμμετοχή σας. Ε, να περάσετε ένα εξαιρετικό βράδυ. Οι ε, ε, συζητήσεις θα συνεχίσουν αύριο στις 9 η ώρα το πρωί. Διακόπτεται η συνεδρία.